Okay, colleagues, we're a bit late starting, um, but I'm glad colleagues are here because we're going to discuss something. Συνάδελφοι, ξεκινάμε λίγο αργά, αλλά θα συζητήσουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι ε, η, ο υποσυτισμός στη Σομαλία, την Ιγερία και χώρες της ε, Αφρικής. Θα ήθελα να δούμε λίγο κάποια πράγματα για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ακούσω γιατί σε κάποιες χώρες, ας πούμε με το Ελνίνιο, έχουμε λιμό και σε άλλες όχι. Πώς το καταφέρνουν, υπάρχουν μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτές, υπάρχουν πολίτες που αναρωτιούνται στην αρχή του 21ου αιώνα πώς έχουμε αυτές τις ε, εικόνες, υπάρχουν σειράξεις μεν, αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει το κλίμα και άλλα τέτοια ζητήματα. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε λοιπόν είναι τι γίνεται για να απαλληλθούν οι άμεσες ανάγκες, τι λείπει ακόμα και αν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό. Αν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, τι κάναμε λάθος, τι ε, υπάρχει τώρα ως εναλλακτική. Έχουμε το θέμα της ανθεκτικότητας, τα ζητήματα που αναφέραμε σήμερα το πρωί και που συζητήσαμε στην Ολομέλεια. Αυτά είναι τα πράγματα που θέλουμε να ε, συζητήσουμε. Έχουμε το, τρεις ε, ε, καλεσμένους, τον Βανσάν Ιμπάν, επικεφαλής της υπηρεσίας OCHA του Ηνωμένου Εθνών, το Γραφείο Σύνδεση τη Βρυξέλλες, Ανδρούλα Καμινάρα, Διευθύντρια για την περιοχή της Αφρικής Ασίας, Λατινική Αμερική, Καραβικής και Ειρηνικού και το Λέοναρτ Μίτζη, επικεφαλής της Περιφερειακής Ανάπτυξης και του της επισητιστικής ασφάλειας. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητοί βουλευτές. Ε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο Σουδάν, την Νοτιοανατολική Νιγηρία και τη Σομαλία. Αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο σημαντικές επισητιστικές κρίσεις ε, της εποχής μας. Πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον λοιμό ή ε, είναι ε, στα πρόθυρα του λοιμού. Μεταξύ αυτών 1,4 εκατομμύρια παιδιά. Πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και έχουμε και εξάρσεις χολέρας πάνω από 20 ε, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν υγιεινή ε, ε, καθαρό νερό και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να εκτοπίζονται είτε εσωτερικά είτε ως πρόσφυγες. Αυτοί που φεύγουν από τα σπίτια τους, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους λόγω σύραξης, πλήττονται περισσότερο από αυτή την κρίση, από, τον, την πείνα, από το λοιμό. Έχουν ε, διαλυθεί ολόκληρες κοινωνίες, ε, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι οικογένειες πάσχουν. Ο λοιμός δεν είναι απλώς θέμα επισητιστικής ασφάλειας. Έχει να κάνει με το πόσο ευάλωτοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, δεν, έχουν τη, οι οποίοι δεν έχουν τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν έχουν ελπίδα τα παιδιά. Δεν πηγαίνουν στο σχολείο παρόλο που αποτελούν το μέλλον των χωρών αυτών. οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, δεν έχουν πλέον τα βασικά, υπάρχει αστάθεια σε όλη την περιφέρεια και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Το νότιμο Σουδάν έχει κηρύξει τοπικό λοιμό. Σομαλία, Ιεμένη και Νιγηρία κινδυνεύουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κρίσεις αυτές τις χώρες είναι παρατεταμένες και περίπλοκες. Υπάρχουν εδώ και χρόνια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παρατεταμένη φύση των σειράξεων η οποία παρατείνει και τις κρίσεις ταυτόχρονα. Όλες αυτές οι χώρες έχουν προβλήματα προσβασιμότητας λόγω ανασφάλειας και κάποιες έχουν και γραφειοκρατία που κοστίζει πολύ και ε, επιδεινώνει τα δεινά των πολιτών. Στη Σομαλία το 1 τρίτο των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από το Αλσαμπάκ, όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Στο Νότιο Σουδάν η χώρα παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου για να είσαι ε, μέλος ε, μιας ανθρωπιστικής αποστολής στην νοτιοανατολική Νιγηρία, όπου το Μπόκο Χαράμ συνεχίζει να κάνει επιθέσεις σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. 700.000 ε, άνθρωποι ε, είναι σε σημεία μη προσβάσιμα και ζουν σε απεγνωσμένες συνθήκες στην Ιεμένη, όπου συνεχίζει η σύραξη ε, και η κρίση υπάρχουν ε, προβλήματα σε περιοχές και λιμάνια που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Πριν από νέα εβδομάδες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να προλάβει αυτή την καταστροφή. Ζήτησε από όλους τους παράγοντες να συνεργαστούν για να σώσουν ζωές, να μειώσουν την ευαλωτότητα και να ε, αυξήσουν την ανθεκτικότητα στα μελλοντικά ε, σοκ, στα μελλοντικά προβλήματα και οι τέσσερις χώρες ήδη ε, επιζητούν ε, βοήθεια σε επίπεδο επισητιστικό. Χρειάζεται λοιπόν ε, μεγάλη κλιμάκωση των δράσεων σε σχέση με το όσα συνέβαιναν πριν γίνει αυτή η έκκληση από τον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σύντομα λοιπόν θα σας δείξω τώρα κάποια βασικά νούμερα. Στο Νότιο Σουδάν εκτιμούμε ότι πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι ζητούν άμεση επιστημιστική βοήθεια. 100.000 από αυτούς βρίσκονται σε δύο επαρχίες που ήδη πάσχουν από λοιμό. Από το Φλεβάρι είμαστε στο 1,2 εκατομμύρια. 300.000 από αυτούς είναι σε τις επαρχίες που πλήττονται περισσότερο. Στη Σομαλία με 3 εκατομμύρια άνθρωπα, ανθρώπους να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους επιστηστικές ανάγκες. Σχεδόν 1 ε, εκατομμύριο παιδιά φαίνεται ότι θα υποσυτιστούν φέτος. Έχουμε επιπλέον την χολέρα και διάρρεια. Στη Σομαλία έχει διπλασιαστεί η αντίδραση από το Φλεβάρι και 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βοήθεια σε επίπεδο επισητιστικό. Στην Ιεμένη έχουμε τη μεγαλύτερη επιστημιστική και κρίση και κρίση ασφαλείας στον κόσμο. 17 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πρόβλημα, 7 εκατομμύρια εξ αυτών ζητούν άμεση επιστημιστική βοήθεια. Μισό εκατομμύριο παιδιά πάσχουν από σοβαρό υποσυτισμό. Εχθές είχαμε στην ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο μια ε, λεπτομερή επισκόπηση της κατάστασης ε, στην νοτιοανατολική στην βορειοανατολική Νιγηρία έχουμε πάλι, πολλά εκατομμύρια ανθρώπους πάλι που ζητούν άμεση επιστημιστική βοήθεια 1,8% ε, εκατομμύρια ε, πάσχουν από αρρώστιες και 4 εκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί κατά της ηλαράς. Οι δωρητές επίσης ε, έχουν δεσμεύσει 26% των άμεσα απαιτούμενων κονδυλίων. Αυτό είναι μια ποσόστοση του ποσού που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό που ονομάζουμε καταστροφή. Σήμερα στην Γενέβη ελπίζουμε ότι η διάσκεψη που γίνεται εκεί ε, θα δώσει τα κονδύλια που θέλουμε, όπως θα γίνει και με τη διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία η ανθεκτικότητα, η αντίσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική. Οι συνάδελφοι θα σας πούν περισσότερα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ευχαριστήσουμε όμως για όσα έχουν γίνει από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη. Και αυτό συμπεριλαμβάνει, εκτός από το λοιμό, την κινητοποίηση των πολιτών, τουλάχιστον σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, όπου στο Βέλγιο, ας πούμε, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε μεγάλη κινητοποίηση. Ο κύριος Ομπράιον επίσης ε, που ήρθε πέρυσι τον Νοέμβρη για να μιλήσει για τη Συρία και άλλες σοβαρές ε, ε, κρίσεις μας έδωσε στη διάθεσή μας 80 εκατομμύρια δολάρια μέσα από το Emergency Response Fund. Οι επιχειρήσεις στις χώρες αυτές ε, φέτος επιζητούσαν 5,8 δις ε, δολάρια, τα 4,4 άμεσα. 1,30 μόνο έχουμε πάρει. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειάζεται να σώσουμε ζωές και πρέπει να το κάνουμε επιγόντως. Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που απαιτούνται. Πρώτον, περισσότερη πολιτική βούληση για να σταματήσουν οι σειράξεις που προκαλούν αυτές τις κρίσης. Πρέπει να σταματήσει η σύραξη, η βία, να εφαρμοστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανθρωπιστικές, γιατί αλλιώς οι ανθρωπιστικές συνθήκες ε, και η πιστιστική ανασφάλεια θα συνεχιστούν, όπως και ο λοιμός και ο ποσιτισμός. Δεύτερον, όλα τα μέρη της σύραξης πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκτυο δίκαιο και να επιτρέπουν στις ανθρωπιστικές αποστολές και όσους εργάζονται σε αυτές να έχουν πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη. Και τα Δύο μέρη πρέπει να τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις. Τρίτον, χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση για να ενισχύσουμε αυτή την αντίδραση και την απάντηση στην κρίση από τους δωρητές, από τις αναπτυξιακές τράπεζες και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Τέταρτον, ζητάμε ένα νέο τρόπο εργασίας μετά από αυτή την κρίση. Δεν είναι αρκετός αυτός που έχουμε για να μειώσουμε τους κινδύνους και την ευαλωτότητα. Χρειάζεται ταυτόχρονη κλιμάκωση των δράσεων και προγραμματισμός. Για να, γίνει, για να αυτό χρειάζεται να ανεχτούμε περισσότερους ε, κινδύνους, περισσότερο ρίσκο, να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο προσαρμοστικοί. Το Μάρτιο τα Ηνωμένα ε, Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας, ανέφερε τη δημιουργία μιας επιτροπής για το λοιμό και την πρόληψή του ε, στις τέσσερις αυτές χώρες με την παρουσία της Παγκόσμιας Τράπεζας οι συνάδελφοι και της ΕΦΚΟ ε, συνεργάστηκαν και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Πρέπει να σταματήσουμε το λοιμό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για τη συνεχή υποστήριξή σας πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στο προσωπικό που θα φέρνει όλα αυτά τα δύσκολα εγχειρήματα σε πέρα. Τώρα η Αντούρα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω στέλνοντας κάποια βασικά μηνύματα για τους λοιμούς στις τέσσερις αυτές χώρες και θα πω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωση στη συνέχεια. Καταρχάς, ο, ο, η λέξη λοιμός, αυτός καθεαυτός, παρόλο που έχει κηρυχθεί επισήμως ένα μέρος της περιοχής στο νότιο Σουδάν, στη χώρα αυτή, σε άλλες χώρες λέμε ότι είμαστε πολύ κοντά, πλησιάζει, μιλούμε για επικείμενο λοιμό και στις τέσσερις περιπτώσεις. Είναι, ο κόσμος ε, δεν έχει δει τέτοια κρίση από το 1945 μέχρι σήμερα και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη λοιμό στα τελευταία έξι χρόνια. Την τελευταία φορά που υπήρξε λοιμός υπήρξε το 2011. Τώρα ξαναχρησιμοποιούμε επισήμως αυτό τον όρο λοιμός και μάλιστα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Στη διάσκεψη που πρόσφατα οργανώσαμε στο περιθώριο της διάσκεψης για τη Συρία κάποιος είπε ότι μπαίνουμε στην τέλεια καταιγίδα και μάλιστα σε τέσσερις ε, τέλειες ε, καταιγίδε παράλληλες που θα κινούνται στις εκάστοτε τέσσερις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πολύ ενεργητική δράση και προσπαθεί ε, να καταπολεμήσει την κατάσταση αυτή σε αυτές τις χώρες και σε αυτές τις περιοχές. Το 2016 έχουμε δώσει 345 εκατομμύριο ευρώ. Δεν θα αναφέρω πάρα πολλά νούμερα, ούτε θα μιλήσω ιδιαίτερως για το χρήμα. Άλλωστε ο Λέοναρτ θα αναφερθεί σε αυτά. Σε γενικές γραμμές θα ήθελα να τονίσω κάποια που έχουν ήδη τονιστεί. Πρώτον, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρώτον, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Δεύτερον, χρειάζομαστε καλύτερη πρόσβαση στον πληγέντα πληθυσμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μιλούμε για περιοχές που δεν ελέγχει εκάστοτε ε, κυβέρνηση ή περιοχές που ελέγχονται από την Πόκο Χαράμε μεταξύ άλλων. Άρα ε, το Διεθνές Δίκαιο για τα ανθρωπαστικά θέματα ε, θέματα και ο ανθρωπιστικός χώρος που θα πρέπει να μας επιτραπεί είναι ζωτική σημασία για να παρέμβουμε και να αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση. Τρίτο σχόλιο που θα ήθελα να διατυπώσω είναι το εξής. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μια αιτία που οφείλεται στον άνθρωπο, ανθρωπογενή αιτία. Δεν λέμε ότι το 100% των αιτιών είναι ανθρωπογενές, ωστόσο ε, πάντοτε υπάρχει μια ανθρωπογενής αιτία πίσω από αυτή την κατάσταση, εν μέρη. Και θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ένας παράγοντας που ευθύνεται, είναι πολύ παραγωγικό το εκάστοτε ζήτημα των, ε, του καθενός από τους τέσσερις λοιμούς που μαστίζουν τις χώρες αυτές. Μιλούμε για μια πλειάδα προβλημάτων που αθρίζονται, που συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο και επιβαρύνουν την κατάσταση αθρηστικά. Και τέταρτον, τελευταίον, ε, πρέπει να αναφέρουμε τις περιφερειακές επιπλοκές. Δηλαδή, ε, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη Σομαλία ή στον Νότιο Σουδάν και τέλος, αυτά που συμβαίνουν εκεί επηρεάζουν την ευρύτερη γειτονία, την ευρύτερη περιοχή και πρέπει κανείς να τα ε, δει υπό αυτή τη σκοπιά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να παρεύει αποτελεσματικά. Δύο λόγια να σας πω για την κάθε χώρα, για την Ιγυρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και παρέχει στήριξη από το 2015 Έχουμε μαζικά εντύν τις προσπάθειές μας έκτοτε. Να μην λησμονούμε όμως ότι πέρσι το καλοκαίρι οι αρχές της Νιγηρίας ήταν πολύ επιφυλακτικές και δεν ήθελαν να παραδεχθούν το μέγεθος της κρίσης της ανθρωπιστικής και της κλιμάκωσής της. Πρόσφατα άλλαξαν στάση και με πολύ θετικό τρόπο οι αρχές της Νιγηρίας, η κυβέρνηση της Νιγηρίας ήταν από τους συν οικοδεσπότες της διάσκεψης όπου υποσχεθήκαμε το 1 τέταρτο της συνολικής βοήθειας που ε, θα προκύψει. Το 1 τέταρτο προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίσημη δέσμευσή της στη σχετική διάσκεψη. Για τη βόρειο-ανατολική Νιγηρία μιλούμε για το σύνολο της περιοχής του Τσάντ. Καμερούν, Νιγηρία, Τσάντ. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό πρόβλημα η βόρειο-ανατολική Νιγηρία. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς, όταν σήμανε για πρώτη φορά το καμπανάκι του συνεγερμού και αναγνωρίστηκε η κατάσταση ως κρίσιμη, τότε πολύ λίγοι ήταν οι εταίροι που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Ε, ήταν και δύσκολες οι πτήσεις. Πάρα πολύ λίγοι ήταν παρόντες. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά. Πάρα πολλές με κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μετακινήσει τους πόρους τους, έχουν στείλει ανθρώπους επιτόπου, αλλάζει η κατάσταση. Η πρόσβαση παραμένει δύσκολη βέβαια. Έχουμε τις πρόσφατα απελευθερωθεί στις περιοχές και στις περιοχές που, έχετε που έχουν απελευθερωθεί πρόσφατα μπαίνουν ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και βλέπουν ότι δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Δεν υπάρχουν καθόλου ούτε σχολεία, ούτε πόροι, ούτε σπόροι, ε, δυνατότητες γεωργικής εκμετάλλευσης, καλλιέργειας, γιατί τα έχουν κάψει όλα προτού τα εγκαταλείψουν. Ε, είναι λοιπόν επίγουσα η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να δράσει κανείς σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε περιόδους βροχών, περιόδους φύτευσης, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Φαίνεται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες και η πιο κρίσιμη και δύσκολη περίοδος θα είναι το καλοκαίρι από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο για τη βορειοανατολική Νιγηρία. Μιλούμε λοιπόν για πολλά και διαφορετικά προβλήματα στην περιοχή της λίμνης του Τσάντ. Ε, πάρα πολλά σημεία είναι σε υποανάπτυξη για πάρα πολλά χρόνια, άρα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και όταν τα χτυπά τα σημεία αυτά και τις περιοχές αυτές η κρίση τα είναι περιοχές που είναι ακόμα πιο ευάλωτες από ό,τι άλλες ή από ό,τι ήταν οι ίδιες στο παρελθόν. Τώρα, έχουμε και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ιγυρία. Πριν από κάποιους μήνες ε, είχαμε βομβαρδισμό σε ένα καταβλισμό προσφύγων, βομβαρδισμό κατά λάθο από το στρατό της Νιγηρίας. Έχουμε δηλαδή και τέτοιου είδους προβλήματα. Μια, ένα περίπλοκο κοκτέιλ μια περίεργη περίπλοκη μίξη των προβλημάτων. Πολύ συχνά οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους όχι μόνο και κυρίως λόγω της Μποκοχαράμ αλλά και λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης της Νιγηρίας να μην ξεχνούμε ότι μέχρι πριν από ένα-ενάμιση χρόνο ε, αυτή η χώρα θεωρείται ως η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική και τη διακηρύσαμε ως τέτοια. Η Νιγηρία μέχρι πριν από ένα-μισή χρόνο δεν άνοικε στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και το επίπεδο της φτώχειας ήταν ε, πολύ χαμηλό. Σίγουρα έχει πληγεί η χώρα αυτή από τις εξαγωγές, από τις τιμές του πετρελαίου που έχουν καταβαραθρωθεί. Ωστόσο, υπάρχει ευθύνη ε, της κυβέρνησης της Νιγηρίας και πρέπει να δει τι το καλύτερο μπορεί να κάνει ε, για τις περιοχές της χώρας που ε, μαστίζονται, διότι η κυβέρνηση της χώρας έχει ίδιους πόρους. Άρα δεν το λέω για να το τονίσω, απλά ήθελα να το θέσω υπόψη σας και έρχομαι τώρα στις άλλες χώρες. Νότιο Σουδάν. Η κατάσταση εδώ είναι τελείως διαφορετική. Αυτή είναι μια καταστροφή αποκλειστικά και μόνο ανθρωπογενής. Ούτως ή άλλως η χώρα ήταν πάρα πολύ φτωχή προηγουμένως. Τα προβλήματα υφίσταντο, υπήρχαν. Όμως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την συνεχιζόμενη σύγκρουση. Δύο εκατομμύρια πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν υπολογίζεται ότι θα έχουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Δύο εκατομμύρια στις γειτονικές χώρες. Άρα ξαφνικά θα πάνε στην Ουγκάντα τη διπλανή η οποία μέχρι πέρσι ε, δεν ήταν και χώρα που μπορούσε να υποδεχθεί ε, τόσο τεράστια νούμερα και αριθμούς προσφύγων. Η Ουγκάντα είναι παριθμόν ένα χώρα που υποδέχεται πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Αφρική και δεν δύναται. Άρα βλέπετε πόσο τεράστιες και σημαντικές είναι οι περιφερειακές επιπλοκές. Το σημαντικό είναι να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο αντιμεχόμενων πλευρών για να πιστούν να σταματήσουν. Τελικά σήμερα είναι σχεδόν σαν να λέμε ότι δεν έχουν κανένα κίνητρο να σταματήσουν, να συγκρούονται. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι του συμφέρει να συνεχίσουν να συγκρούονται για να, προχωρήσει, να, να προωθήσει κάθε πλευρά τη δική της ατζέντα, δυστυχώς. Επομένως, η επικεφαλή των Αποστολών στην Τζούμπα, η ειδική απεσταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέρας της Αφρικής. Έχει εμπλακεί, είναι πάρα πολύ δραστήριοι όλοι αυτοί οι παράγοντες, προσπαθούν να στείλουν αυτά τα μηνύματα, να βρουν ευήκοα όταν και να πείσουν τους ε, συμμετέχοντες να σταματήσουν αυτή τη συνεχιζόμενη καταστροφή. Θα υπάρξει συντονιστική συνεδρίαση μεταξύ των δωρητών και των δρόντων στις 10 και 11 Μαΐου και θα παραστώ εγώ γιατί δεδομένου του μεγέθους της έντασης των ε, πραγμάτων που, συμβαίνει, που συμβαίνουν είναι αθήρητη ανάγκη να ε, συνεργαστούμε, να δουλέψουμε όλοι μαζί, να μην υπάρχουν επικαλύψεις αλλά να μην αφήσουμε και τομείς ακάλυπτους ε, για να αξιοποιήσουμε όλους τους δυνατούς πόρους και αυτός είναι ένας από τους στόχους της συνάντησης στις 10 και 11 Μαΐου. Έρχομαι τώρα στη Σομαλία και εδώ έχουμε ένα, μια βεντάλια προβλημάτων, με ένα μείγμα προβλημάτων. Το 2011 ήταν ο τελευταίος λοιμός στη Σομαλία, μετά από μια χαμένη περίοδο βροχών, 50.000 άνθρωποι πέθαναν το 2012 λόγω αυτού και τώρα έχουμε σύγκρουση επιτόπου, έχουμε ε, απουσία πρόσβασης, έχουμε ξηρασία, έχουμε νέα κυβέρνηση πολλούς και διαφορετικούς δηλαδή παράγοντες που αθρηστικά ε, δημιουργούν αυτό το κίνδυνο. Οι προβλέψεις είναι δυσμενείς. Έχουμε το κακό σενάριο και το χειρότερο σενάριο. Δεν έχουμε καλό σενάριο εκεί. Το κακό σενάριο είναι να υπάρξουν κάποιες βροχές που αναμένονται κατά μέσο όρο ή να είναι κάπως καλύτερες και άρα θα υπάρξει ανάγκη για μαζική αύξηση των κονδυλίων. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι να μην βρέξει και καθόλου, οπότε τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, πολύ χειρότερα για αυτούς και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη αύξησης των κονδυλίων. Με ρωτάτε λοιπόν, τι είναι το σφάλμα, τι θα μπορούσαμε να κάνει διαφορετικά. Ας δούμε τι έγινε με το Ελνίνιο, τι είχε κάνει η Θεοπία, τι είχε κάνει η Κένια τότε. Κοιτάξτε, υπήρξε μαζικότερη κινητοποίηση όλων των ταμείων, όλων των κονδυλίων. Ε, η Κένια έχει ήδη βάλει δικά της χρήματα από το δικό της προϋπολογισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Άρα αυτές είναι οι διαφορές. Θα έπρεπε να είχαμε δρεώσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ε, αυτό το κάναμε εν μέρη για τουλάχιστον να μην μας έρθει ξαφνικό και τώρα ξέρουμε λοιπόν ότι έρχεται αυτός ο λοιμός, είναι, επίκειται και ξέρουμε τι μας περιμένει. Είναι σημαντικό ε, να ε, ε, δουλέψει η κυβέρνηση για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και να μην είναι τόσο ευάλωτη μπροστά στα μελούμενα. Ένα θέμα με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία είναι για παράδειγμα το εξή. Υπάρχει μια πόλη, η Μπαϊντιόα, που στεγάζει 30.000 ανθρώπους. Πολλοί πήγαν εκεί να εγκατασταθούν γιατί κατάλαβαν ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι διάφοροι εταίροι εκεί έχουν εγκατασταθεί και μπορούν να δώσουν βοήθεια. Από το Μογκαντήσου μέχρι αυτή την περιοχή, αυτή την πόλη υπάρχουν 40 σημεία ελέγχου για τα φορτηγά και κάθε φορά ε, ζητείται ένας φόρος εντός εισαγωγικών, ένα χαράτσι, κάθε φορά που περνάει κανείς από τα 40 σημεία εισόδου το ε, φορτηγό και υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα επιτόπου για την ε, παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας και τέλος θα ήθελα να πω ότι είναι η ΕΜΕΝΗ σήμερα γίνεται μια πολύ σημαντική σύσκεψη για το θέμα αυτό στη Γενέβη. Μια διάσκεψη δέσμευσης και υποσχέσεων των δωρητών. Ο Επίτροπος Τηλιανίδης είναι στη Γενέβη αυτή τη στιγμή και έχει πολύ μεγάλες ανακοινώσεις να κάνει εξ ονομάτως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή επιπρόσθετων κονδυλίων για τη χώρα αυτή. Δεν θα σας πω τα νούμερα. Να σας πω όμως ότι για τα παιδιά μόνο μιλούμε για 500.000 παιδιά τα οποία ε, υποσυτίζονται ε, έντονα, ε, πάσχουν από σοβαρό υποσυτισμό. Στην Ιεμένη λοιπόν οι περιφερειακές επιπτώσεις είναι ίσονος σημασία συγκριτικά με τις άλλες τρεις χώρες, ωστόσο η, έλλειψη ισχύω του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της προστασίας των αμάχων πληθυσμών και της υποδομής είναι παντελής η έλλειψη αυτή και άρα η πρόσβαση είναι πολύ μεγάλο ζήτημα εξίσου, η πρόσβαση η δική μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Άρα, αυτά έχω κατά κύριο λόγο να σας πω. Συνοψίζω λέγοντας ότι έχουμε τέσσερις λοιμούς ή επικείμενους λοιμούς και ε, δημιουργούνται οι συνθήκες για την απόλυτη καταιγίδα. Ε, και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με το βέλτιστο δυνατό ε, τρόπο. Ευχαριστώ. and good afternoon. Um, Ευχαριστώ. Έχω ένα σύντομο PowerPoint και μετά θα προσπαθήσω να συμπληρώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι της Σότσα. Αυτό το οποίο βγαίνει από τη συζήτηση αυτή μέχρι τώρα είναι η ανάγκη για ένα νέο παράδειγμα σε επίπεδο συντονισμού. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σε συνεργασία με το JRC και την ΕΚΟ και την FAO και άλλους διεθνείς εταίρους έτσι ώστε να γίνει μια τεχνική διαδικασία, μια τεχνική συζήτηση η οποία οδήγησε στην σφαιρική, στη συνολική έκθεση. Η έκθεση αυτή κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου. Δεν ξέρω, μπορώ να σας δώσω τον σύνδεσμο αν θέλετε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αναλυτική προσπάθεια η οποία έχει γίνει και θα πρέπει να συμπληρωθεί και από μια πολιτική διαδικασία τα θέματα δεν είναι μόνο κλιματολογικά, αλλά και πολιτικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να διευκολύνουμε τον πολιτικό διάλογο και να προωθήσουμε τον συντονισμό. Η τεχνική διαδικασία, για να σας δώσω κάποια αναλυτικά στοιχεία, για κάθε χώρα υπάρχει μία ανάλυση του τι είναι αυτό που επηρεάζει την κρίση. Κλιματολογικό, σαν παράδειγμα αν είναι συνδυασμός διαφορετικών πολιτικών και μη πολιτικών, επιδημιολογικών μορφών επιθέσεων θα έλεγα. Καθορίζουμε επίσης και τις τάσεις και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και τη γεφύρωση των διαφορετικών κατεπηγουσών καταστάσεων. Αυτή είναι η σφαιρική έκθεση, δεν θα μπω στους αριθμούς, έχουν ήδη αναφερθεί. Έχετε την κατάσταση στις τέσσερις χώρες, έχετε τις αιτίε οι οποίες αναφέρθηκαν από τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Αυτό το οποίο εδώ είναι νέο, είναι το ξεκάθαρο αίτημα και μια σαφής απάντηση σε πολιτικό επίπεδο. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και τα Ηνωμένα Έθνη, να έχουν πιο στρατηγική αντιμετώπιση, να έχουν μια σφαιρική καλύψη και να καλύπτουν το σύνολο του πολιτικού πεδίου. Να συντονίζουν επίσης καλύτερα ε, τα οικονομικά μέσα, είτε τα DCI, είτε το EDF, είτε τα ε, καταπιστεύματα. Πέρυσι 540 εκατομμύρια ε, κινητοποιήθηκαν για να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που έθεσε το Ελνίνιο. Το πώς δουλεύει τώρα η πολιτική διαδικασία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε το πεδίο στο οποίο θα γίνει η πολιτική συζήτηση και να βελτιώσουμε ε, τον, ε, το επίπεδο συντονισμού σφαιρικά συνολικά. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα λοιπόν στις κρίσεις οι οποίες υπάρχουν στον τομέα των τροφίμων όταν μάλιστα δημιουργούνται από ε, αστάθεια και δημιουργούν συγκρούσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να δημιουργήσουμε ένα θερμόμετρο για το σύστημα early warning, εγκαίρις προειδοποίησης, να δούμε ποια είναι τα λεγόμενα hot spot, να δούμε και ε, βραχυπρόθεσμα τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε μέσω πρόθεσμα. Ένα παράδειγμα στην Ιγυρία. Για την Ιγυρία έχουμε κινητοποιήσει όχι μόνο χρήματα από την ΕΚΟ, αλλά έχουμε δημιουργήσει και το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα στα 130 εκατομμύρια, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα. Μιλάμε πολύ για αντοχή και ανθεκτικότητα. Θα πρέπει λοιπόν και με τη δική σας στήριξη να υποστηρίξουμε τη γεωργική παραγωγή. Μιλήσαμε για τις διακοιμάνσεις των τιμών και για τα καύσιμα που παράγει η χώρα, όπως επίσης και το, τις τιμές, την αύξηση της τιμές των προϊόντων, την απότομη αύξηση στις τιμές των διαφόρων προϊόντων και αγαθών επίσης βελτίωση της αγοράς απασχόλησης, αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και ανθεκτικότητα στον τομέα της υπαίθρου. Το πώς θα δημιουργήσουμε τώρα την ανθεκτικότητα αυτή και σε προληπτικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με περιοχές οι οποίες εκτίθενται συχνά σε καταστροφές, Επίσης το θέμα της ανθεκτικότητας στις κλιματολογικές αλλαγές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλήματα στον τομέα του εισίδρευσης. ενδεικτικά εθνικά προγράμματα, αγαθά δημόσια, αναχώρα, δίκτυα επικοινωνίας και αύξηση του επίπεδου προετοιμασίας, έγκαιρη προειδοποίηση για τυφώνες. This is the case of, of in Western Africa. Περιπτώσεις λειψιδρίας επίσης. Τίθεται επίσης και το θέμα της διαφοροποίησης της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε επίσης και τις υποδομές, κάλυψη των ζημιών μετά από την παραγωγή, και αύξηση της ανθεκτικότητας στους τομείς τους οποίους οι ίδιες χώρες δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Αναφερθήκαμε στην Κένια και την Αιθιοπία. Όταν υπάρχει μια σαφής στρατηγική για την ανάπτυξη της υπαίθρου με εθνική χρηματοδότηση, προτεραιότητες στον τομέα της διασφάλισης της παροχής τροφίμων σε εθνικό επίπεδο, μειώνονται οι κίνδυνοι και είναι λιγότερο ευάλωτες οι χώρες οι οποίες ε, έχουν πάρει τα μέτρα σε σχέση με τις προτεραιότητές τους. Τώρα το πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα σε άλλους τομείς όπου έχουμε ανοιχτές σειράξεις σαν παράδειγμα. Κέντρο Δημοκρατία. Εμπλέκεται και το FAO και ε, τοπικές ε, οργανώσεις. Ε, διανομή τροφίμων ad hoc σε συγκεκριμένες χώρες και στη Σομαλία μεταφορές ποσοτήτων τροφίμων σε περιοχές όπως ενίση του πράσινου ακροτηρίου. Όπως επίσης και η λογική της αντιμετώπισης του θέματος της αλυσίδας αξιών σε χώρες όπως η ακτή του ελεφαντοστού <coughs> και προσπάθειες αποκατάστασης, αποζημίες που μπορούν να αποκαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο την καθημερινότητα. Συνεργαζόμαστε εδώ με την ΕΚΟ και με τις εξωτερικές υπηρεσίες, όπως και με την υπηρεσία που έχει την έδρα της στη Ρώμη, έτσι ώστε και μέσα από τη σφαιρική έκθεση και με τις περιοδικές ενημερώσεις να δώσουμε κάποιες απαντήσεις που να είναι καλές σε επίπεδο λειτουργικό και να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό διάλογο βελτιώνοντας όπως είπα την ανθεκτικότητα της ζωής των ανθρώπων στις γεωργικές περιοχές, στις περιοχές της Υπέθρου. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε τις παρουσιάσεις σας. Ο Γκουερέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τους τρεις εισηγητές που μας παρουσίασαν τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των τεσσάρων αυτών χωρών. Ήδη έχουμε επισημάνει ότι είμαστε μέσω τεσσάρων τέλειων απόλυτων καταιγίδων οι οποίες εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμυρία οι οποίες φέρνουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε μια κατάσταση απόλυτης ανέχειας και αδυναμίας επιβίωσης. Το σίγουρο είναι ότι η πρώτερη κατάσταση από την δήλωση της Άμπρουνα ήταν πολύ σημαντική. Ήδη είχαμε εκατομμύρια εκτοπισμένους, ανθρώπους που έχουν δυσκολία να έχουν πρόσβαση στη σύντηση, ε, συνθήκη ζωής απολύτως δυσχερής. Επίσης ε, είναι βέβαιο αυτό που υπόθηκε. Ότι δηλαδή, όταν εξαρτάται η ζωή κάποιου από το αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει και ότι το αποδεχόμαστε αυτό ως κακό σενάριο γιατί μπορεί να υπάρχει το χειρότερο σενάριο του να μην βρέξει καθόλου κιόλας. Όταν ε, το δέχεται κανείς αυτό, ουσιαστικά διαπιστώνει απουσία ανθεκτικότητας, αδυναμία αντοχής όλων αυτών των περιοχών, οι οποίες δεν δίνανται να αντιμετωπίσουν αυτές τις επίγουσες καταστάσεις. Εξού και σήμερα το πρωί σε αυτή την Επιτροπή ψηφίσαμε τη θέση μας ως Επιτροπή ΝΤΕΒΕ για την ανακοίνωση που έχει να κάνει με την αντοχή, την ανθεκτικότητα, τον τρόπο με τον οποίο βοηθάει κανείς ώστε ο, ο ενδεής να μην εξαρτάται από τα φυσικά φαινόμενα κατά 100% αλλά να μπορεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες περιπτώσεις. Και μετά από τους τρεις συζητητές αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα είναι το εξής. Αυτό που πυροδοτεί τις κρίσεις ε, ε, είναι ανθρωπογενές. Υπάρχει μια αιτία ανθρωπογενής. Δεν είναι μόνο μια αιτία που έχει να κάνει με φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι ότι επειδή ήρθε φέτος το Ελνίνιο θα υπάρχει ξηρασία ή λειψίδρια κτλ. Μιλούμε για χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση πάρα πολλά χρόνια, που εκτοπίζουν ανθρώπους που ε, υψώνουν εμπόδια στην βασική ανθρώπινη ε, συναλλαγή και δραστηριότητα που καταστρατηγούν ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Άρα, ε, οφείλουμε να προβληματιστούμε και να πούμε ότι μαζί με τη μεγαλύτερη οικονομική προσπάθεια πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για πολιτική συνομιλία, συνδιαλλαγή, για να μετριάσουμε τις ένοπλες συγκρούσεις και για να επιτύχουμε να επιτρέπεται η πρόσβαση των δρόντων σε ανθρωπιστικό επίπεδο στις ζώνες σύγκρουσης. Άρα, πώς θα συμβάλλουμε στο να μειώσουμε τις συγκρούσεις και πώς θα διασφαλίσουμε ότι στις περιοχές συγκρούσεων θα φτάσει η βοήθεια στους πληθυσμούς που το, το χρειάζονται, που την χρειάζονται. Αυτά τα δύο είναι αμοιώς πολιτικές δράσεις. Δεν είναι δράσεις που απαιτούν οικονομικούς πόρους. Είναι πολιτικές δράσεις, πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις λάβει στο σύνολό της και οι σχετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για διάφορους λόγους έχουν κάτι να πούν και έχουν, θέλουν να είναι συνομιλητές με τις χώρες όπου σημειώνονται αυτές οι κρίσεις. Τέλος, θέλω να υποβάλω δύο ερωτήματα. Υπόθηκε ότι στη διάσκεψη που γίνεται σήμερα στη Γενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και ο Επίτροπος Τηλιανίδης θα δεσμευτεί για ενίσχυση και αύξηση της βοήθειας. Έχετε πληροφορίες. Τι θα κάνουν οι άλλοι δωρητές. Ποιες είναι οι άλλες προοπτικές για την ουσιαστική αύξηση της οικονομικής συνεισφοράς για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Και αν δεν απατώμε, υπόθηκε ότι υπάρχουν 7-8 χώρες της Ένωσης που απάντησαν στις δεσμεύσεις που ε, αναλήφθηκαν. Δηλαδή, θα μπορούσαμε ως Επιτροπή να υιοθετήσουμε κάποια πρωτοβουλία, να υποβάλουμε κάποιο ερώτημα, τα έχουμε κάνει βέβαια αυτά σε περασμένες ολομέλειες συνόδους ολομελιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να απαιτήσουμε, να απαιτήσουμε από τις χώρες της Ένωσης που κάποια στιγμή είχαν δεσμευτεί να ε, κομίσουν κεφάλαια για να βοηθήσουν την, ε, το μετριασμό αυτής της κρίσης, να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε οι σχετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και δεν θέλω να ε, μιλήσω ονομαστικά, αλλά στις χώρες που αναφέρατε δεν αναφέρατε τη δική μου χώρα. Η Ισπανία είναι τέταρτη οικονομική δύναμη στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ και αν η κυβέρνησή μας ήταν προοδευτική, σίγουρα θα συνέβαλε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο στο μετριασμό των ε, κρίσεων και των, ε, της δυστυχίας αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μαρία Χόιμπουκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις πολλές καλές και σημαντικές πληροφορίες. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για τη γρήγορη απάντηση, αντίδραση και τις άμεσες ε, Θα ήθελα καταρχάς λοιπόν να ευχαριστήσω τη Γενική ε, Διεύθυνση ΕΚΟ για τις άμεσες πληρωμές σε αυτήν την ε, ε, κρίση την επισητιστική. Περίμενα να ακούσετε τη διερμηνία. Νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην Ευρώπη σε αυτά τα θέματα και ξέρουμε ότι στο Σαχέλ και στην Αφρική το θέμα αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Εμείς ε, παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια και σημαντική βοήθεια, όμως ταυτόχρονα η Ευρώπη πρέπει να αναρωτηθεί ποιοι είναι οι λόγοι. Γιατί φτάνουμε σε αυτά τα διέξοδα σε επίπεδο επισητιστικό οι αναλυτές και εδώ στην αίθουσα έχουμε μερικούς ε, λένε ότι δεν έχουμε μόνο τις φυσικές καταστροφές όπως το Ελνίνιο αλλά ε, δεν είναι μόνο αυτές, είναι και οι πολιτικές καταστροφές που παίζουν ένα ρόλο. Αναφέρθηκε ότι οι άνθρωποι προκαλούν αυτές τις κρίσεις. Είναι ανθρωπογενείς. Στην Σομαλία, στο Σουδάν έχουμε ε, τους ηθήνοντες ε, της διεφθαρμένες κυβερνήσεις οι οποίες δεν φροντίζουν το λαό τους στην Αιθιοπία. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό, μια τεράστια χώρα στην οποία υπάρχει λειψιδρία, ε, αλλά δεν υπάρχει αυτό που ε, θα θέλαμε, η λογοδοσία στη δημοκρατία και η διεθνής κοινότητα ε, απλώς παρακολουθεί πώς αφήνουν το λαό τους να πεινάει. Δεν υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη στη γεωργία ε, παραβλέπεται η γεωργία και από τη γεωργία προέρχονται οι τροφές, τα τρόφιμα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν αν η Κομισιόν στη συνεργασία της στον τομέα της γεωργίας είναι ικανοποιημένη. Ε, γίνονται όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να φτάσουν τα τρόφιμα στους ανθρώπους, να τραφεί ο πληθυσμός. Είστε ικανοποιημένοι με τη συνεργασία, πώς λειτουργεί και ως Κομισιόν πώς μπορείτε να έχετε επιρροή στις χώρες έτσι ώστε να αποφύγουμε στα επόμενα πέντε χρόνια να μιλάμε για τις επόμενες επισητιστικές καταστροφές επειδή παραβλέψαμε πράγματα που είχαν προβλεφθεί. Η δυνατότητα ανθεκτικότητας, ε, η αντίσταση είναι μια πολιτική ε, πραγματικότητα που παραγράψατε. Τι γίνεται όμως στις ίδιες τις χώρες ποιες είναι οι οικολογικές μέθοδοι που ε, χρησιμοποιούνται, που θα πρέπει να προωθήσουμε έτσι ώστε να ε, μπορούμε να αντισταθούμε. Να υπάρχει ανθεκτικότητα και οι βιομηχανικές μέθοδοι. Επίσης, θα με ενδιέφερε ε, να ακούσω, κύριε Μίτσι, πόσο ρεαλιστική είναι η επιτυχία της Sacrifice αυτή την κρίση στις χώρες. Έχει συνεισφέρει ώστε να μην έχουμε στο μέλλον άλλες ε, επιστημιστικές ε, κρίσεις ή παρά την συνεργασία που υπάρχει ε, θα έχουμε πράγματα σαν αυτά που βλέπουμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Ήθελα μέσα στα πλαίσια του More for More ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες προέλευσης, χώρες ε, διαμετακόμισης για τους ε, μετανάστες, είτε πρόκειται για διδεκτατορίες, απολυταρχικά καθεστώτα, είτε δημοκρατίες, αν, να δούμε αν παίρνουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων του Γιούνκερ. Επίσης, αυτές οι δραματικές επενδύσεις μέσω της Agrify. Πώς συμβάλλουν σε όλα αυτά. Σε χώρες όπως το Σουδάν, με τους ιδιώτες επενδυτές ε, ε, μπορεί κανείς να φτάσει στη Γεωργία. Φτάνει εκεί. Ε, το χρήμα είναι η εξουσία που υποστηρίζεται μόνο. Και επίσης από τη νέα συμμαχία για την επιστηστική ασφάλεια ξέρουμε ποια είναι η επίδραση των επενδυτών αυτών. Δεν φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, στις ντόπιε επιχειρήσεις, αλλά στους μεγάλους ομίλους και ακούμε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση για τη νέα αυτή συμμαχία και για τις ε, διμερείς συνομιλίες που είχατε περίπου για τρεις ε, μήνες περίπου και θα ήθελα να μάθω γραπτός κάποια πράγματα για αυτή τη νέα συμμαχία γιατί δεν πήραμε τίποτα σε σχέση με αυτά που γίνονται, για τον τρόπο, για την ποιότητα των όσων έχουν επιτευχθεί θα χαρώ λοιπόν πολύ αν μπορούσα και γραπτός να έχω αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Okay, thanks, Maria. A lot of questions there about... Ευχαριστούμε Μαρία. Πολλές ερωτήσεις για πολλά πράγματα. Αλλά όπως και να έχει ε, είναι ένα θέμα η ανθεκτικότητα και ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα ζητήματα. Νόρμπερτ, είσαι ο επόμενος και μετά ο Ζωακή Μισέλα. Ε, ευχαριστώ. Από τη δική μου πλευρά και πάλι ευχαριστώ πολύ για την πολύ άσχημη αυτή αναφορά για την κατάσταση των ανθρωπογενών αυτών κρίσεων όπως υπόθηκε των πολιτικών κρίσεων. Το ερώτημα τώρα είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά η βοήθεια ε, θα πρέπει να αυξηθεί. Αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πολύ καλά Έχω μία ερώτηση σχετικά με την Ιγυρία, γιατί σε αυτά τα κράτη, τα τέσσερα που αναφέρατε, η Νιγηρία φαίνεται να διαφέρει λίγο σε σχέση με τα άλλα, με τον εμφύλιο πόλεμο. Ε, ε, ο εμφύλιος με το Μπόκο Χαράμ δεν είναι κάτι μικρό. Ε, επίσης έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι και φαίνεται ότι έχουμε μια αλλαγή κυβέρνηση στην Ιγυρία, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση η οποία ήρθε με τη βία και θέλει να περιορίσει τον Μπόκο Χαράμ και την επέκτασή του, την προέλασή του. Έχουμε κάποιες δυνάμεις στα, όρια, στα σύνορα με το Τσάτ, το Καμερούν, τον Ήγυρα και στα ε, βόρειο-δυτικά ε, της ε, Νιγηρίας έχουμε και εκπροσώπους των Joint Military Forces όπου υπάρχουν συνομιλίες με αυτούς και μπόρεσαν πιστικά να επηρεάσουν ώστε τον Μπόκο Χαράμ να μην έχει πλέον τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα στην καταστολή και στους ε, ε, μηχανισμούς καταστολής που χρησιμοποιεί. Στην Νιγηρία η, η όδευση δεν είναι θετική σε αντίθεση με τις άλλες τρεις χώρες τα το τελευταίο διάστημα. Η πορεία δεν έχει πάρει μια θετική τροπή. Είναι μια χώρα η οποία είναι ε, σχετικά ελεύθερη ε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ε, πολλά θέματα πετρελαίου όπως πριν τι γίνεται με την Ιγυρία λοιπόν ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τις άλλες χώρες ο Γιώχημ Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές για τις πληροφορίες. Νομίζω ότι θα συνταχθώ με τον Μάρκους για αυτά που είπε και με όλους τους προλαλήσαντες σε σχέση με το γεγονός ότι η κατάσταση στις τέσσερις αυτές χώρες αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια έχει πολιτικές ε, ε, διαστάσεις και δεν πρέπει διπλωματικά να μιλούμε πλέον. Θα πρέπει ε, με τις ανθρωπιστικές δράσεις από το εξωτερικό μεν να δραστηριοποιηθούμε αλλά αυτό δεν βοηθά πλέον επαρκώς θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους εκτοπισμένους οι οποίοι εσωτερικά ή εκτός των συνόρων μετατοπίζονται, εκτοπίζονται για να αποφύγουν τα δεινά. Ε, όπως είπε και ο Νόρμπερτ ε, για την Ιγυρία, η σύραξη με τον Μπόκο Χαράμ είναι πολύ καιρό. Είχαμε μεγάλες ελπίδες για τον ε, πρόεδρο Εν μέρη μπόρεσε να τις εκπληρώσει, αλλά δυστυχώς εδώ και πολλές εβδομάδες είναι ε, άρρωστος και δεν μπορεί να ε, ανταποκριθεί στα καθηκοντά του. Είναι στο Λονδίνο για να γιατρευτεί, για θεραπεία. Ε, στο μεταξύ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την καλλιεργήσιμη υγιή και πολλά ζητήματα που οδηγούν σε σειράξεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε τι βαθμό ένα κράτος ε, και αυτοί που το κυβερνούν ε, λογοδοτούν και πρέπει να λογοδοτήσουν. Στο νότιο Σουτάν, εκεί πέρα, οι warlords που ζουν από τον ε, πόλεμο τα πάνε καλά και στο Ναϊρόμπι είχαμε τις εκλογές στην στο μεταξύ είχαμε εγκλήματα πολέμα, πολέμου από τις αουδαραβικές δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις Έχουμε λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα ίδια πράγματα. Η διεθνής κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη τελικά θα πρέπει να υψώσει το ανάστημά της και να ονοματίσει τους υπεύθυνους. Εκεί που πολιτικά είχαμε παρέμβει με κυρώσεις, ε, είχαμε κάποιες δυνατότητες ε, να κάνουμε μια αλλαγή. Ε, εδώ έχουμε ανθρώπους σε, μιζέρια, σε ανέχεια. Είναι πολλές οι χώρες που πάσχουν. Είχα πολλές φορές τη δυνατότητα σε κάποιες από αυτές τις χώρες να πάω και όταν υπάρχει κάποια σχετική ειρήνη και τάξη και πολιτική ε, σταθερότητα και μια διακυβέρνηση μπορεί να συτιστεί το διπλάσιο ποσοστό πληθυσμού. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να υποστηρίξουμε τις μοντέρνες μεθόδους π.χ. Ε, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υγείας, υποσυτισμού ε, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να παρεύουμε πριν αναλάβουν βιβλικές διαστάσεις όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο ότι όποτε μπορούμε θα πρέπει να παρέμβουμε, να φτάσουμε σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, αλλά να μην έχουμε την ε, παρέστηση ότι με αυτά που εμείς εδώ δίνουμε, ότι θα μπορέσουμε στο μεταξύ να ε, ανταποκριθούμε πλήρως ε, στο πρόβλημα, να το λύσουμε, ας πούμε, σε αυτό, αυτά που γίνονται στην Αραβική Χερσόνησο. Είναι πολιτικά ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της ε, δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν γίνουν τα σωστά βήματα, οι σωστές ε, δράσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αναλάβουν και αυτά δράση και όχι απλώς να μιλούν. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγινε μια αίτηση για τις ε, εξαγωγές ε, όπλων στο Νότιο Σουδάν να σταματήσουν. Ε, δεν υπάρχει πλέον πλειοψηφία για αυτήν. Νομίζω ότι σε αυτό φταίει η διεθνής κοινότητα. Έχει συνυπευθυνότητα για αυτό το θέμα. Είναι κράτη αυτά τα οποία ζουν μαζικά από την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να δούμε και ποια είναι η δική μας ευθύνη σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Ευχαριστώ. Ανελίτς. Επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε μόλις ο κύριος Θέλεο. Υπάρχουν προτάσεις από πλευρά σας για το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δράσει. βλέποντας ακριβώς όλες αυτές τις πολιτικές συγκυρίες τις οποίες αναφερθήκατε. Έχετε κάποια στοιχεία στην έρευνά σας έτσι ώστε να μας δώσετε κάποιες κατευθύνσεις θα έλεγα για να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε. Λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος λέει η πρόεδρος. Όχι. Η Σεσίλ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που προηγήθηκε για την έλλειψη των τροφίμων και για τις τέσσερις αυτές χώρες στις οποίες αναφερθήκατε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λίγο κάποια βασικά θέματα τα οποία οδήγησαν, θέλετε, στην κρισιμότητα αυτής της κατάστασης και της έλλειψης τροφίμων όπως επίσης και της ξηρασίας που επικρατεί στις χώρες αυτές. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της φυσικής καταστροφής από τη μία, στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε πολιτικά και οικονομικά. Τίθεται όμως και το πολιτικό θέμα. Έχουμε να κάνουμε σε πολλές από αυτές τις χώρες, σε όλες τις χώρες αυτές, δεν υπάρχει θα έλεγα μία πολιτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου το πρώτο πράγμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι οι διαδικασίες ειρήνευσης. Εκεί που έχουμε κάνει τέτοιες προσπάθειες και εκεί που έχουμε υπογράψει συμφωνίες ε, με χώρες που δεν υπάρχει ειρήνη, χώρες τις οποίες δεν γνωρίζουμε αν τα χρήματα αυτά φτάσουν τελικά στον πληθυσμό, φοβάμαι ότι δεν βοηθούμε τις χώρες αυτές έτσι ώστε να καταφέρουν να ξεφύγουν από τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Ένα τμήμα των χρημάτων αυτών φτάνει στον πληθυσμό, τα υπόλοιπα μένουν στις τσέπες των κυβερνώντων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στις πολιτικές ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού. Το δεύτερο θέμα είναι η ενίσχυση των κρατικών δομών. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία, η Εμένη, και σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις ε, ε, ζήτησα να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε καλύτερα το τι γίνεται στην Ιεμένη. Οι περισσότεροι Ιεμενίτες πηγαίνουν στο Τζιμπουτί και στις υπόλοιπες χώρες ε, της περιοχής. Εκεί δεν βοηθούνται, δεν καταφέρνουν λοιπόν να ζήσουν στην Ιεμένη, καταλήγουν στο κέρας της Αφρικής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα τους βοηθήσουμε να ξεφύγουν από την κρίση αυτή. Όταν το κράτος δεν υπάρχει, όταν είναι εξασθενημένο, δεν υπάρχουν δομές οι οποίες να μπορέσουν να κάνουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Και σκέφτομαι τα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να βοηθήσουν στην σωστή διακυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Χωρίς την ενίσχυση των κρατικών δομών δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε σε ποιον θα πάνε. Και το τελευταίο είναι η λεγόμενη ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα μας επιτρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε άμεσα με τους τοπικούς πληθυσμούς. Υπάρχει μια κάποια μορφή αποκεντρωμένη συνεργασίας για την ανάπτυξη. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε απευθείας στους πληθυσμούς ξεπερνώντας το φαινόμενο της συγκέντρωσης των εξουσιών, την κεντρική εξουσία. Όταν πολλές από τις μορφές της βοήθειας περνούν από την κεντρική κυβέρνηση, σπάνια φτάνουν ε, στην υπόλοιπη χώρα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει αναπεριφέρεια, μπορεί να γίνει αναπόλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς με σωστό τρόπο κλείνω αναφερόμενοι στα τοπικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και την κατάρτιση των νέων. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην βελτίωση της ανθεκτικότητας, έτσι ώστε οι ίδιοι κάτοικοι να μπορέσουν να βγουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και οι γυναίκες, σαν παράδειγμα, και οι νέοι έχουν τις δυνατότητες, αλλά δεν έχουν τις δομές που θα τους συνοδεύσουν δεν έχουν τους συνεταιρισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να βελτιώσουν την αντοχή τους. Ξεκινήσαμε με ένα μέλος και τώρα έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είναι τόσο σημαντική η συζήτηση, ε, είναι πολλές οι ερωτήσεις, δεν ξέρω με ποιον θα ξεκινήσουμε. Παρακαλώ να είστε συντομότατοι γιατί έχουμε ε, καθυστερήσει τουλάχιστον κατά μισή ώρα. Κάποιες από τις ερωτήσεις έχουν σχέση με ανθρωπιστική βοήθεια και με μακροπρόθεσμες διαδικασίες ανάπτυξης. Εγώ παρουσιάζοντας την κρίση είπα ότι συνεργαστήκαμε στενά με την ΤΕΦΚΟ εντοπίσαμε 14 χώρες στα πλαίσια του προγράμματος αυτού που ακολουθούμε και τις συμπεριλάβαμε στον κατάλογο. Οι υποσχέσεις τώρα ε, για την ιεμένη συνάντηση γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι και ο Επίτροπος Τηλιανίδης θα δώσει υποσχέσεις για περαιτέρω μορφές χρηματοδότησης και από ΕΚΟ και από ΝΤΕΦΚΟ. Και αυτό οφείλεται και στο ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά για τις κρίσεις αυτές. Σε σχέση τώρα με το σύνολο των χρημάτων τα οποία δαπανώνται, το σύνολο των χρημάτων τα οποία προτείνονται. Εμείς εξετάσαμε σε σχέση με το ODA ε, τη στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και βλέπουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνεται γενικά, αλλά στην Αφρική ε, μειώνεται ειδικά. Αυξάνεται το τελικό ποσό, αλλά στις περιοχές τις οποίες αναφερόμαστε, σε τρεις από τις χώρες αυτές, μειώνεται. Για την Αφρική λοιπόν. Υπάρχει συνεπώς ένα θέμα εδώ, το θέμα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα υποσχόμεθα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε. για το τι συμβαίνει στην Ιγυρία και αν τα πράγματα βελτιώνονται ή ου. Υπάρχει αύξηση των βομβιστών αυτοκτονίας και έχουμε και περιπτώσεις δυστυχώς 7-8 ετών ανθρώπων που ανατινάσσονται, παιδιών που ανατινάσσονται. Όταν το παιδί φτάνει μέσα στην ομάδα των ανθρώπων, κάποιος με τηλεχειριστήριο το τεινάζει στον αέρα μαζί με τους παρόντες γύρω του. Είναι απρόβλεπτη πολύ η κατάσταση δυστυχώς. Είναι συνεχώς όλο και πιο περίπλοκοι η όροι με τους οποίους εμείς εργαζόμεθα στην Ιγυρία. Οι πολιτικές επίσης συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Τέθηκε το ερώτημα τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια των ΑΚΕ και των συμφωνιών και της κοινοβουλευτικής συνέλευσης μπορεί να συζητηθεί ότι κάποιες, κάποια από τα προβλήματα αυτά μπορεί να οφείλονται στην εγκατάλειψη κάποιων περιοχών των χωρών αυτών στην εγκατάλειψη κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών παραγόντων ή κάποιων μειονοτήτων συνολικότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορείτε να σας απασχολήσει. Στην περίπτωση της Νιγηρίας κάτι τέτοιο είναι σαφές. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικά θέματα που χειροτερεύουν την κατάσταση. Θα συμφωνήσω μαζί σας επίσης ότι η πολιτική αστάθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά κάθε χώρα βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Στη Σομαλία έχουμε μια νέα κυβέρνηση, είναι ένα θετικό βήμα, πρώτο βήμα, αλλά είναι μια μακρά, μακρά, μακρά διαδικασία πριν καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική πολιτική κατάσταση. Λοιπόν, αυτά έτσι ώστε να έχουν χρόνο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να απαντήσω στην κυρία Χόιμπουκ. Συνεργασία για γεωργικά ζητήματα, για ε, επισητιστική επάρκεια, ασφάλεια διατροφής και ούτω καθεξής. Σήμερα η διαδικασία είναι διαφορετική από την Λακουίλα, όπου είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση κονδυλίων. Η κατάσταση σήμερα είναι κάπως διαφορετική. Η αρχιτεκτονική δομή της οργάνωσης των δωρητών είναι τελείως διαφορετική από αυτή που υπήρχε πριν από 7 ως 10 χρόνια. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όσο τον περισσότερου πόρου και να προωθήσουμε μια ατζέντα που θα βάζει τη γεωργία και την επιστημιστική ασφάλεια και επάρκεια στο πυρήνα ε, των ανησυχιών μας, αλλά έχουμε και κίνδυνο διάδοσης και μετάδοσης. Δηλαδή, αν δεν έχουμε σταθερότητα σε μια χώρα, αυτό ε, μεταφέρεται και στις άλλες και γι' αυτό μίλησε για το αποθεματικό τροφίμων της ECOWAS, της ECOWAS που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής. Ναι, χρειαζόμαστε πιο συνολική προσέγγιση. Δεν μπορεί κανείς να έχει ε, διατροφική ασφάλεια, επάρκεια, επισητιστική επάρκεια, χωρίς να έχει μια σωστή προσέγγιση για το εμπόριο και να μην υπάρχει εμπορική ολοκλήρωση των σχέσεων ε, της, εντός ε, της ίδιας περιοχής τουλάχιστον. και θα πρέπει να αναλαφθεί ε, δράση όταν η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και δεν αποδίδεται μόνο σε φυσικές καταστροφές. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλα τα είδη επενδύσεων, δημόσιες επενδύσεις αλλά και ιδιωτικές που συμπεριλαμβάνουν εκφύσιους πιο πολλούς συμμετέχοντες. Ξέρετε ότι προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να ε, δεσμεύσουμε τους ιδιώτες επιχειρηματίες για να αναλάβουν καινοτόμο δράση. Και αυτό θα απασχολήσει ε, την πρωτοβουλία του G7 που θα εξεδιπλωθεί τις επόμενες εβδομάδες, τα τέλη Μαΐου. Και θα υπάρχουν και τα θέματα επάρκειας, ε, γεωργίας και το καθεξής. Θα πάμε και στο Βερολίνο, όπου και η κυβέρνηση προσπαθεί να κινητοποιήσει τη χάρτα του Βερολίνου για την απασχόληση στην Ήπεθρο και για το πώς απασχολούμε τους νέους στην Ήπεθρο και το πώς ενισχύουμε τις υποδομές, πώς έχουμε επιχειρηματικά μοντέλα και τα εφαρμόζουμε στην Ήπεθρο. Προσπαθούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλες τις προσεγγίσεις, όλες τις, όλους τους τρόπους δράσης και σε επίπεδο G7 και σε επίπεδο G20 για να έχουμε πιο συντονισμένη δράση η χρήση γης, η κατοχή της γης, η ύπαρξη γης είναι κάτι το απαραίτητο για να υπάρχει σταθερότητα. Και θα μιλήσουμε για την 50η ε, επέτειο των εθελούσεων κατευθυντήριων γραμμών. Θα, στη Ρώμη τον Οκτώβριο θα έχουμε παρουσίαση ειδικών περιπτωσιολογικών μελετών εκεί όπου υπάρχουν success story, ιστορίες επιτυχίας, εκεί όπου έχουμε ενεργητική αγροτική πολιτική, κρατεή, ισχυρή, συμπεριληπτική, κεντρική διοίκηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, ε, επιχειρηματικά μοντέλα, εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Αυτά όταν υπάρχουν έχουμε επιτυχίες και προσπαθούμε να έχουμε κεντρική προσέγγιση όμως, όταν οι ανώτατες πολιτικές υποδομές δεν δουλεύουν, όταν δεν υπάρχει ενδοϊπουργικό συντονισμός, ενδοϊπηρεσιακός, ο Υπουργός Γεωργίας να συνομιλεί με τον Υπουργό Οικονομικών, να συνομιλεί με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όταν δεν υπάρχουν αυτά δεν έχουμε ίδια εμπλοκή, ίδια εμπιστοσύνη, ίδιο θετικό αντίκτυπο. Εκεί όπου δίδονται δυνατότητες στον Υπουργό Γεωργίας και έχουμε αποκεντρωμένη δράση, η επιτυχία είναι πιο εγγυημένη και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα όπου η κατάσταση αλλάζει, όπου ο ρόλος των οργανώσεων των αγροτών ε, είναι σημαντικός παρόλο που αυτές βρίσκονται σε ευρυκό ακόμα στάδιο. Και σαφέστατα προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να ε, συμβάλλουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για την αποτελεσματικότητα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό για όλους, για τις δωρήτριες χώρες βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε με αυτές τις επιτροπές, με τη συνάντηση με τους αρμοδίους από το Γενικό Γραμματέα στην Ηνωμένα Έθνη και με άλλους, είναι να ε, αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, να ε, λύσουμε τα σημεία στα οποία σημειώνεται κυκλοφοριακή συμφόρηση, να κινητοποιήσουμε ανθρώπους και χρήματα. Αυτή είναι η βασική στόχη. Ε, μιλήσατε για τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα. Είναι ένας τρόπος να γίνουν όλα αυτά και συμφωνούμε και πράγματι πρέπει να υπάρξει ε, μια τέτοια απάντηση, αλλά υπάρχουν και άλλες. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα συντονίσουμε σε αυτή τη συνέργεια μεταξύ δωρητών και ε, λιπτών της βοήθειας. Μιλούμε επίσης για τα εργαλεία χρηματοδότησης. Προσπαθούμε τα χρήματα να φτάσουν ώστε να τον πιο κοντά στις κοινότητες αυτές καθεαυτές. Άρα σας διαβεβαιούμε ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστούν όλα αυτά εφικτά και δυνατά. Νομίζω ότι όλοι είπαμε τι μπορεί να γίνει και ήδη το κάνετε εσείς αυτό. Την τελευταία χρονιά υπήρξε ένας αριθμός ψηφισμάτων που ανέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπήρξε πίεση που ασκήσατε εσείς στις χώρες μέλη, ε, στις χώρες που πρέπει να δράσουν. Το σημαντικό είναι να δώσουμε ένα τέλος στη σύγκρουση και ε, όταν τελειώνει η σύγκρουση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ε, ε, μένουν οι άνθρωποι χωρίς την προστασία της μίας από τις δύο ένοπλες ομάδες και γι' αυτό πρέπει να έρθουμε εμείς να καλύψουμε αυτό το κενό και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι το 2011 όταν κηρύχθηκε ο λοιμός στη Σομαλία είχαμε ήδη 200.000 θανάτους πριν τον κηρύξουμε, μέχρι να τον κηρύξουμε. Εμείς δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί. Ξέρουμε τι χρειάζεται, ξέρουμε ότι συνεχώς ζητούμε, και για, συνεχώς ζητούμε χρήματα και είναι δύσκολο, αλλά πράγματι τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ώστε να το περισσότερο η πολιτική πίεση μπορείτε να ασκήσετε και αυτές οι τέσσερι χώρε να ξέρετε είναι πολύ διαφορετικές. Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, τα ίδια προβλήματα, αλλά είναι διαφορετικές, άρα διαφορετικό είναι ο τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε κάθε μία. Και Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευθεί ότι θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και βασιζόμαστε σε αυτές τις χώρες και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ε, δυσάρεστη και θλιβερή η εικόνα που μας περιγράφεται. Τις εικόνες αυτές τις έχουμε δει και στην τηλεόραση πάρα πολλά χρόνια τώρα και βλέπουμε ότι θα τις ξαναδούμε δυστυχώς. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ε, κάποιες αιτίες είναι ανθρωπογενείς, άλλες αιτίες έχουν να κάνουν με το κλίμα, με το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας και οτιδήποτε χρειάζεστε να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Ε, μιλήσαμε για τις χώρες ΑΚΕ και ίσως πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί ε, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης με τις χώρες ΑΚΕ να τους ε, ρωτήσουμε πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ιγυρία, τι γίνεται με την Μπόκο Χαράμ. Ας ε, το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ για να μην παραπεταχθεί, να μην χαθεί αυτό. Τον Ιούνιο δεν είναι η συνάντηση με τι χώρες ΑΚΕ, σωστά. Άρα... Ήδη το πράξαμε. Πολύ συχνά, ξέρετε, όμως οι εταίροι μας από τις πληγήσεις χώρες Ε, δεν θέλω να το συζητήσουν. Ξέρετε, εγώ ήμουν από μια χώρα, από μια περιοχή όπου είχαμε μείωση της, ε, και πολύ μεγάλη παρακμή της βιομηχανικής παραγωγής και όταν έγινε λόγος να μπει η περιοχή μου στις περιοχές στόχου 1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι, ε, κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι πολύ κακό αλλά όταν είσαι φτωχό είναι καλύτερα να μπει στο στόχο 1 και να λάβεις όλη τη βοήθεια που χρειάζεσαι ακόμα και αν αυτό ε, δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί γιατί είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε του ομιλητέ θερμά. Um, Προχωρούμε λοιπόν στην εξέταση του επόμενου σημείου της ημερήσιας διάταξης. Θα ε, έρθουν οι επόμενοι προσκεκλημένοι. Θα χρειαστούμε ένα-δυο λεπτά ε, μέχρι να ε, έρθουν οι νέοι προσκεκλημένοι να λάβουν τις θέσεις τους, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα αμέσως. Okay, colleagues. Um, moving on to item 17. Ωραία, συναδελφοί. Περνάμε στο 17 που είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο γιατί έχουμε μία μελέτη, έχουμε επίσης και μία έκθεση από την κυρία Χιμένεθ Μπεσρίλ Γι' αυτό το θέμα. Πρόκειται για τον συνεχώ συρρυκνούμενο χώρο της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε πολλούς εταίρους από χώρες που μας λένε ότι υπήρχε αυτή η στιγμή που επεκτηνόταν η δημοκρατία και γινόταν εκλογές. Τώρα όμως φαίνεται ότι υπάρχει μία καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ε, μειώνονται σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η Τερέζα Χιμένες Βεθερίλη είναι η συγγήτριά μου η Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια ε, σχετιζόμενη επιτροπή και υπάρχει και μια συζήτηση που θα ξεκινήσει γιατί έχουμε μια μελέτη. Έχουμε το πεδίο και την έκταση του προβλήματος. Έχουμε τρεις ε, ε, ομιλητές, τον εισηγητή ο οποίος είναι στο, εφέλος στο Carnegie Europe, κανείς ωραία από την ACT Alliance ε, και η κυρία Μπεν Τόπαΐς από την DG DEFCO για τις, ε, που είναι υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά σε αυτό το τομέα. Έχω μία συνάντηση στις 5, ο κύριος Βάριον θα αναλάβει στις 5 ως ε, πρόεδρος και του δίνω το τώρα αυτό το αδύνατο να μειώσει το χρόνο της συνεδρίασης. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση μία ώρα, πρέπει να τελειώσει στο χρόνο, πάνω στο χρόνο που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα όμως και χρειαζόμαστε ε, μεγάλη προσοχή. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιάνξ. Θα μας δώσει την άποψή του για τον διεθνικό συνεκρούμενο χώρο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεσή μου περιγράφει το πώς οι περιορισμοί στην κοινωνία των πολιτών στον κόσμο επιδεινώνονται σε μεγάλο βαθμό και περιγράφει πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πρόβλημα και πώς εντατικοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει θέσει σε εφαρμογή μια εντυπωσιακή σειρά νέων ε, πρωτοβουλειών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ ήθελα να εξετάσω σε ποιο βαθμό αυτή η πολύ καλή δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια να συνεχιστεί. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πιο, ακόμα πιο αποτελεσματική την απάντησή της στο πρόβλημα. Ένα από τα βασικά ζητήματα της έκθεσης έχει άμεση σχέση με την επιτροπή σας. Στο μέλλον η πρόκληση είναι η κοινωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ε, για, τις, ε, για να μπορούν οι πόροι της αναπτυξιακής βοήθειας να χρησιμοποιούνται πλήρως ώστε να έχουμε μια στρατηγική απάντηση στο πρόβλημα του συρρυκνούμενου χώρου. Μέχρι τώρα υπάρχει το αίσθημα ότι αυτό το πρόβλημα γενικά έχει επηρεάσει την κοινωνία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει να κάνει με ένα επιλεγμένο αριθμό ξεκάθαρα προβεβλημένων ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλέον το πράγμα δεν είναι έτσι. Έχουμε ένα ευρύ διαρθρωτικό πρόβλημα που πλήττει την κοινωνία των πολιτών και την αναπτυξιακή εργασία και να θέτει προσκόμματα στις πολιτικές της αναπτυξιακής σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι η αναπτυξιακή κοινότητα πρέπει να ενσωματώσει αυτό το θέμα στον τρόπο που σχεδιάζει τις πολιτικές της. Κοιτάζουμε λοιπόν τι έχει γίνει ως τώρα, πόσο καλές ήταν οι πολιτικές, πώς έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία τους. Υπάρχουν πολλές καλές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχουν γίνει για να προστατευτούν οι ακτιβιστές οι οποίοι γνωρίζουμε πόσο κινδυνεύουν σήμερα. Φαίνεται επίσης πόσο πολλά περισσότερα πράγματα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για να δημιουργήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις οργανώσεις των, ε, της κοινωνίας των πολιτών ώστε να αντιμετωπίσουν ε, τους ε, βάναυσους αυτούς περιορισμούς με τους οποίους είναι αντιμέτωπες και κατά πώς η DCI και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν γενικά προβλήματα όπως το, η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεστε αυτό ε, θα βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά η πρόκληση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία εντατικοποιεί και βελτιώνει τη δική της απάντηση, όμως οι κυβερνήσεις στον κόσμο γίνονται όλο και πιο μαχτηρές και σκληρές στις τακτικές που χρησιμοποιούν ενάντια στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα σήμερα. Παρόλα αυτά και παρόλο που το κάνουμε παραμένουμε ε, καθυστερημένοι γιατί το πράγμα τελικά οδηγεί σε επιδείνωση και όχι σε βελτίωση. Ένα από τα ερωτήματα που υποχρεωνόμαστε να θέσουμε είναι το εξής. Σε κάποιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να διατηρήσει το επίκεντρο στην αναπτυξιακή πολιτική, αλλά το έκανε με τέτοιο τρόπο που παραγνώρισε τις τους πολιτικούς στόχους και υποβάθμισε την πολιτική εμπλοκή. Κάτι που οδήγησε στο πρόβλημα αυτό του συρρυκνούμενου χώρου, όπως σε χώρες, ε, σε χώρες όπως την Αιθιοπία, τον Μπαγκλαντές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να διατηρήσει παραγωγική ε, εστίαση στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα να διατηρήσει την πολιτική πρόσφυση σε αυτό το πρόβλημα. Ε, πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά να γίνει προμηθής και όχι επιμηθής. Πρέπει περισσότερες, ε, περισσότεροι πόροι να πάνε πιο αποτελεσματικά στους ακτιβιστές, όμως πρέπει να γίνουν πράγματα ώστε να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και οι οργανισμοί και οι οργανώσεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις τακτικές των καθεστώτων πριν τα προβλήματα πλήξουν τις ίδιες. Είναι μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ πολιτικής και ανάπτυξης για να μπορέσουμε η αναπτυξιακή συνεργασία στις χώρες του κόσμου να παραμείνει στο προσκήνιο και να μην προσδένεται στο άρμα των ε, πολιταρχικών καθεστώτων για να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές οι μη ε, στις χώρες τους. Είναι δύσκολη ισορροπία αυτή. Ένα που πρέπει να γίνει ίσως στο μέλλον είναι να σκεφτούμε τι είδους άμες, έμεσες μορφές ε, ρεσιμότητας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά. Βλέπουμε ότι Όλο και περισσότερο το πρόβλημα πλήττει όχι μόνο ένα μικρό αριθμό περασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μειώνει το χώρο και για την παραγωγική ανάπτυξη αναπτυξιακών έργων. Το ερώτημα είναι πότε αρχίζει αυτό να γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πώς θα αναπτύξουμε την πολιτική πίεση που πρέπει να ασκήσουμε στα ιδιαίτερα συγκρουσιακά καθεστώτα και ειδικά για τους ε, αναπτυξιακούς παράγοντες στο πεδίο να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουν να χτίσουν συνασπισμούς. Ε, η πάταξη αυτής της συρρήκνωσης θα υπάρξει όταν έχουμε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των ακτιβιστών, της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων, όταν ολόκληρη η κοινωνία κινητοποιηθεί κατά των ολένα ε, και αυξανόμενων περιορισμών έναντι της ε, κοινωνίας των πολιτών. Για να καταλήξω εδώ, να πω ότι στο τέλος της έκθεσης έχουμε πάνω από 20 συγκεκριμένες συστάσεις για πολιτικές. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς να αναφέρω δύο για να τελειώσω. Στο μέλλον, ένα που πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα είναι να υποστηρίξει διάφορες μορφές οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι μορφές ε, θα πρέπει ίσως να είναι λιγότερο ευάλωτες και επιδεκτικές ε, σε, τέτοιες, ε, σε τέτοιους περιορισμούς που τα καθεστώτα κινητοποίησαν εναντίον τους. Ήδη γίνεται κάποια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό αναφέρομαι στην έκθεση έτσι, θα πρέπει βασικά στο σύστημα να γίνουμε λίγο πιο ευέλικτοι, πιο ρευστοί έτσι ώστε να έχουμε μια πολιτική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συρρήκνωσης του χώρου. Και τέλος να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλους διεθνείς παίκτες θα πρέπει να δημιουργήσει μια αφήγηση η οποία θα μιλά περισσότερο για τη σημασία ανάπτυξης των ελεύθερων ε, κοινωνιών της ε, κοινωνίας των πολιών, να πολιτών. Να τα συνδέσουμε όλα αυτά με τους στόχους της χιλιετίας, ε, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην αγγίξουμε μόνο αυτούς τους ακτιβιστές που τα καθεστώτα προσδιορίζουν ως δυτικόφιλους, θα πρέπει να προωθήσουμε διάφορες πολιτικές σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή σκέφτεται να αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική αφήγηση για τη συρρήκνωση του χώρου. Αυτό το στοιχείο στην ουσία θα δείξει πώς οι χώρες ε, που δίνουν πλήρως ε, την αυτονομία στην κοινωνία των πολιτών μπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τις αναπτυξιακούς στόχους. Ευχαριστούμε πολύ για την επισκόπηση. Είναι πολλά από αυτά που πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με τις χώρες που έχουν τα λιγότερα προβλήματα, ποια είναι η γενικότερη τάση. Βλέπουμε τις τάσεις σε διάφορες χώρες που δεν είναι και πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες. λογικά θα πρέπει να έχετε πάρει και τη μελέτη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Καρίν Σορέ από την Act Alliance είναι οργάνωση των ε, εκκλησιών ε, και των οργανώσεων πίστης που προωθούν την ανάπτυξη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονόματος και της Concord και της Civil Society Europe. Η κοινωνία των πολιτών είναι στην ουσία μία μορφή συνεργασίας των πολιτών προς το κοινό καλό, προς το κοινό όφελος. Είναι μία θεμελιώδης ελευθερία, είναι επίσης μία δυνατότητα οικοδόμησης της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Η συνεργασία είναι απαραίτητη για να υπάρξει αλλαγή. Μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι θα έλεγα βασικό χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας που βοηθά την ευημερία όλων των κοινωνικών κατηγοριών εκεί όπου αυτό χρειάζεται. Ένας μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων στον κόσμο φοβάται ότι θα ελεγχθεί και γι' αυτό καταστέλει και ποινικοποιεί την δραστηριότητα της οργάνωσης των πολιτών, οργανώσεων των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι θέλουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα τα πολιτικά των πληθυσμών. Αυτοί οι οποίοι υφίστανται τις διακρίσεις όπως οι μειονότητες αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες για να επηρεάσουν την λήψη ε, των αποφάσεων. Μειώνεται ο χώρος και οι δυνατότητες τις οποίες έχουν για να ακουστούν. Είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς ότι κυρίως οι γυναίκες αυτή η μείωση του χώρου έκφρασης δημιουργεί περισσότερες απειλές εκτός από την αύξηση του κινδύνου σύλληψης ή εξαφάνισης τίθεται και το θέμα του βιασμού και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Επίσης, συκοφαντικές ε, εκστρατείες εις βάρος των γυναικών και γι' αυτό το θέμα της ανταμετώπισης του μειούμενου συνεχώς χώρου δράσης είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την, τις κοινωνίες των χωρών αυτών. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν λοιπόν για να σταματήσει να μειώνεται ο χώρος αυτός και στα Ηνωμένα Έθνη ε, και σε σχέση με τις ευθύνες που έχει ο ιδιωτικός τομέας δίδοντας σαν παράδειγμα μεγαλύτερο βάρος στον στόχο 16 της Ατζέντα 2030 και στον δημοκρατικό χώρο που την περιβάλλει. Είναι σημαντικό όμως πως ε, η εσωτερική και εξωτερική δράση της Ένωσης ε, να λειτουργεί με συνεκτικό τρόπο. Η προστασία της κοινωνίας πολιτών πρέπει να είναι χαρακτηριστικό όλων των πολιτικών όπως της ασφάλειας, του εμπορίου και της μετανάστευσης. Δεν μπορεί η Ένωση να ασχολείται με θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα ή στη Ρωσία, αλλά να μην παίρνει ε, μέτρα όταν συμβαίνουν προβλήματα στα κράτη-μέλη. Σαν παράδειγμα, ο νόμος για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και που βρίσκεται συζήτηση στην Ουγγρική Βουλή ή και οι τελευταίες εξελίξεις στην Πολωνία. Ε, υπάρχει το Civicus που παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και υπάρχουν επίσης ε, και ε, κάποιες μελέτες πρόσφατες από τη Civil Society Europe. Η χρηματοδότηση αυτών των τρόπων παρακολούθησης της συρρήκνωσης του χώρου μέσα στον οποίο ζουν οι οργανώσεις των πολιτών είναι βασική μας αποστολή. Δυστυχώς τα τελευταία μέτρα δημιουργούν προβλήματα χρηματοδότησης και περιορισμούς χρηματοδότησης σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυστυχώς ε, ένα σημείο επίθεσης και ένα κακό μήνυμα από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί με τον κύριο Γιάνγκς πιστεύουμε ότι απαιτείται να υπάρξει μια διπλή αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, συνδυάζοντας τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών και των επιμέρους εθνικών προγραμμάτων στις διάφορες χώρες σε επίπεδο συντονισμού των δωρητών και σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει και να ενισχύσει την στήριξή του σε οργανώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οργανώσεις γυναικών, οργανώσεις ΛΟΑΤ, οργανώσεις ε, ε, αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, θρησκευτικές μειονότητες, ειρηνιστές, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, συνδικάτα, ε, ομάδες προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της γης, οργανώσεις ηθαγενών και γενικότερα πιο παραδοσιακές μορφές κοινωνικών και ανθρωπιστικών εταίρων που αντιμετωπίζουν το θέμα του συνεχώς μειούμενου χώρου δράσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κατάλληλοι και ευέλικτοι τρόποι στήριξης της πρωτοβουλίας στον τομέα της αύξησης των δυνατοτήτων, από κοινού κατάρτισης, έρευνας, προώθησης ιδεών και αρχών, παρακολούθησης και ελέγχου, εποπτείας κτλ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε εθνικό. Μια πρόσφατη μελέτη η οποία συνετάχθη από την Concord με 400 μη κυβερνητικέ οργανώσεις από όλο τον κόσμο δείχνει ότι οι αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωση μπορεί να παίξουν έναν θετικό ρόλο στα πλαίσια του διαφθρωτικού διαλόγου στο εσωτερικό της κοινωνίας των πολιτών, στον τομέα των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναπτυξιακών δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν και θα πρέπει η πολιτική ε, δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την προστασία και την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύουμε ότι είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει ανεξαρτησία της κοινωνίας των πολιτών και ε, να μην εφαρμόζουν απλά οι οργανώσεις αυτές ε, τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίσημο επίπεδο. Να πω ότι και στον, στον τομέα των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, πρέπει να υπάρχει έλεγχος του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών. είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, ε, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος, η βοήθεια η αναπτυξιακή, για να προωθηθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, σας έκανα να σταματήσετε νωρίτερα. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε με εκπροσώπους ε, των τοπικών αρχών, έχουμε αυτή την δυνατότητα τώρα. Έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία των Πολιτών σε ε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και εγώ ίδια θα πρέπει άλλωστε να φύγω γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερο που είμαι εδώ σήμερα και η έκθεση αυτή έρχεται σε μια πολύ επίκαιρη, επίκαιρη χρονική ε, συγκυρία. Έχει να κάνει με το χώρο που συρρυκνούνται για τις οργανώσεις της οργανωμένης ε, κοινωνίας των πολιτών. Τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες ε, και μία από αυτές είναι το υπερηραίωσα κατάσταση, το ευρύτερο περιβάλλον για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους μας. Δεύτερος στόχος της ανακοίνωσης είναι ε, να βοηθήσει έτσι ώστε οι ΜΚΟ να συμβάλλουν στην εκάστοτε χώρα αλλά και στις διεθνείς διαδικασίες. Τρίτη προτεραιότητα είναι να ε, αυξήσουν τις δυνατότητές τους, να μπορούν να ε, λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Όλα αυτά είναι ε, αλληλοσυνδεδεμένα. Μιλούμε για τη διαμόρφωση των όρων και των περιστάσεων έτσι ώστε η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να είναι παράγωνα διακυβέρνησης, διαχείρισης και ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και καλώς έχουμε αυτή τη συζήτηση ε, και συμπληρώνει τα πεπραγμένα του Ιδρύματος Κάρνεκη με την έκθεσή του. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω δύο-τρεις διαφάνειες που συμπεριλαμβάνουν τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να εξάγει μετά από το τετραετές αυτό έργο. Το 2012 αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε μαζί με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Δεν δίνουμε στήριξη με βάση συγκεκριμένα project, αλλά τη στηρίζουμε σε επίπεδο ε, δημοκρατικό, σε επίπεδο διαχείρισης και διακυβέρνησης, συμμετοχή στα κοινά. Υπ' αυτή την έννοια βλέπετε ότι με το πρόγραμμα εξωτερικών σχέσεων αυξήσαμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, πηγαίνει στους αποδέκτες μέσω της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Η αύξηση ήταν κατά 12%. Δύο δις ευρώ δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρόνο στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στηρίζει φορείς και τέτοιου συλλόγους και οργανώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ είναι ο κύριος δωρητή στη τοπική ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και τρίτος δωρητής παγκοσμίως ε, στη συνολική ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια γιατί δείχνει πώς προτιθέμεθα να δράσουμε επί τόπου. Έχουμε λοιπόν κάποιες βασικές αριθμητικές σχέσεις, κάποια νούμερα που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 15% του παγκοσμίου ΑΕΠ, ωστόσο εκπροσωπεί το, 5%, το 55% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και τα 2 τρίτα της βοήθειας που δίδονται στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που εδρεύει στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή στην τοπική κοινωνία το 72% που λαμβάνει εν συνόλο το λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτή την διαφάνεια βλέπετε τη στήριξη στην τοπική οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Είμαστε οι πρώτοι στους πέντε πρώτους και πέρα από τη στήριξη για ε, την ανάπτυξη δυνατοτήτων σε βάθος χρόνου, στόχος είναι να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών να συμβάλλει για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης και της πολιτικής ατζέντας για το 2030. Στηρίζουμε τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ της τοπικής οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και της ευρωπαϊκής οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ε, φαίνονται ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Βραχυπρόθεσμα θέλουμε να προστατεύσουμε τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έγκαιρη παρέμβαση, να διατηρήσουμε τις ροές, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να λειτουργούν στις πιο δυσχερείς και δύσκολες καταστάσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το νομικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε την αντοχή, την ανθεκτικότητα, να καλλιεργήσουμε θετική στάση έναντι της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και ε, να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν καλύτερα στις διεθνείς διαδικασίες. Ε, για να ολοκληρώσω, ελπίζω ότι δεν έχω ξεπεράσει το χρόνο που μου έχετε δώσει. Πρέπει να πω ότι προσπάθησα να σας κάνω μια μικρή επισκόπηση της έκθεσης, τι έχει γίνει από το 2012 μέχρι και σήμερα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένθερμος υποστηρικτής της οργανωμένης κοινωνίας των παλιτών σε όλο τον κόσμο και τις πολιτικές δεσμεύσεις τις μεταφράζει σε συγκεκριμένες πράξεις και έτσι ε, χαράσει και σημειώνει, κάνει τη διαφορά επί τόπου. Είναι περίπλοκη η κατάσταση, το γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουμε το, το πρόβλημα του χώρου που συρρυκνούνται συνεχώς σήμερα στις χώρες Αυτέ αυτές για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σωστά την έκθεση του Ιδρύματος Κάρνεγκη και πολλά άλλα που έχω να πω για την έκθεση, αλλά έχετε τα σημεία αναφοράς για την έκθεση που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα 18 Απριλίου και βρίσκεται διαθέσιμη διαδικτυακά. Μπορείτε να τη διαβάσετε και με χαρά θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Στρέφουμε τώρα προς τα μέλη της Επιτροπής μας για να τους δώσω το λόγο. Η Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλη είναι η συγγήτρια και η πρώτη ομιλήτρια. Μην ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι δύσκολο το όνομά μου. Δυσκολεύεστε να το προφέρετε, αλλά ε, σε όλους συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή για την μελέτη αυτή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις παρουσιάσεις που κάνατε. Συμφωνούμε μαζί σας σαν Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε στενές σχέσεις. Έχουμε τους ίδιους στόχους και θέλω να ευχαριστήσω και αυτά τα οποία είπε, για αυτά τα οποία είπε την κυρία Σοέτ όπως και την κυρία Ροσάριο Βέντο για τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Όπως επίσης και τις σχέσεις μας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους. Είναι σαφές ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη της κάθε χώρας, για τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. η κοινωνία των πολιτών ε, γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε χώρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό διάλογο ο οποίος απαιτείται. Είναι σαφές ότι όπως είπαν οι ομιλητές και συμφωνείτε μαζί σας υπάρχει μια κάποια αύξηση της καταστολής και του χώρου λειτουργίας, μείωσης του χώρου λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών. και γι' αυτό έχει σημασία η έκθεση αυτή έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο χώρος καταστολής της δραστηριότητας της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας της κοινωνίας των πολιτών και γι' αυτό θα πρέπει να εμβαθύνουμε εμείς ε, τις διαδικασίες επεξεργασία μιας πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές. Να συγχαρώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όπως επίσης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει για την βελτίωση των συνθήκων με τις οποίες, κάτω από τις οποίες λειτουργεί, ε, λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών στις χώρες υποανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και στον τομέα των ανεπτυξιακό. Έχει να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι πυλώνας μιας ισχυρής και ισότιμης κοινωνίας, μιας ισχυρής, ε, μια ισχυρή ε, κοινωνία των πολιτών είναι εγγύηση για την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών και ιδιαίτερα στις χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται από πολιτικές, από τη φτώχεια, από τον πόλεμο και όταν υπάρχει υψηλή ε, θα έλεγα πολιτική αστάθεια τότε ε, η κοινωνία των πολιτών ε, πρέπει να έχει την ελευθερία και να ασκήσει τα δικαιώματά της με ειρηνικό τρόπο μέσα σε ένα πλαίσιο και μια ατμόσφαιρα σταθερότητας και ασφάλειας αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν, να προσδώσουμε χώρους ελευθερίας και ε, δημοκρατίας έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να βελτιώσει την δράση της και εδώ θα πρέπει και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να τονώσει τις ε, ε, δυνατότητες συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα μαζί της. Υποστηρίζουμε λοιπόν και τη συμπερίληψη των μειονοτήτων στις λεγόμενες εύθραυστες ευάλωτες ομάδες. Θέλουμε να υπάρξει μια βελτίωση ε, της ε, λειτουργίας ε, της κοινωνίας των πολιτών, μια σωστή δυνατότητα εποπτείας της κοινωνίας των πολιτών, της λειτουργίας της εποπτείας των πολιτών και ιδιαίτερα είναι σαφές ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες μειούται ο χώρος δράσης της κοινωνίας των πολιτών και εμείς θα πρέπει να προσθέσουμε, να προσπαθήσουμε στις χώρες αυτές να κάνουμε το αντίθετο, να βελτιώσουμε τους όρους λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεών της και να διευρύνουμε το χώρο αυτό. Εμείς έχουμε ένα ρόλο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ ισχυρό οικονομικά, αλλά δεν έχουμε έναν ισχυρό αντίστοιχα πολιτικό ρόλο. Και δεν μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την οικονομική επιρροή. Αυτό το οποίο συνέβη στο Λίβανο είναι σαφές. Βλέπουμε όμως ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται στη Συρία και βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες συνδιαλέγονται για την ειρήνευση της περιοχής στις χώρες αυτές δεν περιλαμβάνεται παρά την οικονομική της ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν μένει πάρα πολλά να γίνουν. στα μέσα Μαΐου θα είναι δημόσια, θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες η έκθεση αυτή λοιπόν. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31 Μαΐου και η παρουσίαση επίσημη θα γίνει στις 27 Μαΐου. Yes, thank you. I have uh, three requests for, for the floor. The first... Έχουν ζητήσει τρεις το λόγο. Χόιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, πληροφορίες. Καταρχάς, να αναφερθώ στις ε, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Να πω ότι έχετε ε, με πολύ αδρά χρώματα περιγράψει το τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι δομές που πρέπει να διασφαλιστούν. Παρ' όλα αυτά, ε, ανησυχώ και αναρωτιέμαι για πόσο καιρό η δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα είναι κομμάτι της αναπτυξιακής μας πολιτικής, γιατί είναι αυτονόητο ότι από την στιγμή που ε, οι, εσωτερι... Υπουργοί Εσωτερικών έχουν αναλάβει αυτή την ε, πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της μετανάστευσης, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο πολιτικός ε, διάλογος με τις χώρες εταίρους έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Έχουμε άλλα ερωτήματα και το θέμα της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνουν λιγότερης προσοχής. Ε, τίθεται το θέμα εάν προσέχουμε με ποιον συνεργαζόμαστε. Και είναι και δικαιολογημένη η ερώτηση αν δούμε την μετανάστευση που πρέπει να μειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με δικτατορίες στο Σουδάν, στην Ερυθρέα. Είναι λίγο ε, κοντόφθαλμη αυτή η πολιτική. Ε, νομιμοποιούμε μια συνεργασία με αποτελεταρχικά καθεστώτα που καταστέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα παραβιάζουν και με αυτόν τον τρόπο τα νομιμοποιούμε. Η συνεργασία λοιπόν με αυτές τις απολυταρχικές κυβερνήσεις στην ουσία ε, μειώνει τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών να δράσει και ε, το κάνει αυτό χωρίς να έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Ε, θεωρώ επίσης ότι είναι καλό που στη μελέτη σας ε, αναφέρεστε ακριβώς για αυτό, σε αυτό το θέμα και προτείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δει ε, ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις ε, αυτής της ε, ρεαλιστικής προσέγγισης και ξεκάθαρα με αυτή την συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας στην κοινωνία των πολιτών έχουμε μια εικόνα και επίσης τολμάτε και να θίξετε το θέμα της αιρεσιμότητας Υπάρχουν συστάσεις για αιρεσιμότητα σε χώρες όπου υποστηρίζεται η κοινωνία των ε, πολιτών, ε, να τους δώσουμε δηλαδή more for more. Σε αυτή την περίπτωση η προστασία της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι που θεωρώ ότι με αξιοπρόσεκτο τρόπο προωθείται. Και επίσης ε, και αυτό το more for more στα θέματα της μετανάστευσης, ε, πώς το βλέπουμε, ε, θα το πάμε και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι κάνετε εσείς όταν έχουμε μια συνεργασία για τη μετανάστευση που έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σταματάμε τα κονδύλια προς αυτά τα κράτη, Α, τα συνεχίζουμε. Ε, πώς αντιμετωπίζονται ε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους μετανάστες και επίσης αναφερθήκατε σε κάτι ε, που και εγώ θέλω να αναφέρω, ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο και στο κλίμα των καιρών είναι η χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Έτσι να το πάω λίγο παραπέρα, να πω ότι το σχέδιο της έκθεσης του ΕΛΚ στην ουσία κάνει επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πεδίο χειρισμών της κοινωνίας των πολιτών. Δεν το περιλάβαμε καθόλου στην Επιτροπή μας αυτό το θέμα. Δεν δώσαμε σημασία και υπάρχει μια ε, μαζική κριτική Ε, η έκθεση αυτή πραγματικά είναι λίγο έτσι αμφισβητήσιμη και θα έλεγα ότι πρέπει να την επεξεργαστούμε πολύ ε, για να μπορέσουμε να έχουμε τελικά μια έκθεση σωστή. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Φρουντζούλικα, δεν είδαμε ότι ζητήσατε το λόγο. Έπρεπε να ήσασταν ο πρώτος. Ζητώ συγγνώμη, θα είστε ο δεύτερος. Δεν είναι και τόσο σημαντικό. Η ομάδα μου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά και πάντοτε είναι καλύτερα να μιλά πρώτα μια κυρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο συρρυκνούμενος χώρος, το φαινόμενο αυτό ε, που αφορά στην κοινωνία των πολιτών, επιδεινώνεται συνεχώς. Η παγκόσμια πάταξη της κοινωνίας, των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει βαθύνει και επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 100 κυβερνήσεις έχουν περάσει περιοριστικούς νόμους για τις διαδικασίες των, της κοινωνίας των πολιτών και χρησιμοποιούν επίσημες και ανεπίσημες τακτικές για να θέσουν σε μειονεκτική θέση αυτές τις οργανώσεις. Οι περιορισμοί στην κοινωνία των πολιτών εντατικοποιούνται σε μη δημοκρατικές, αλλά δυστυχώς και σε δημοκρατικές χώρες. Και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακόμα και σκοτώνονται από κάποιες κυβερνήσεις είναι σε αριθμό ρεκόρ στον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει την στρατηγική της για το συρρυκνούμενο χώρο ε, πιο έχουμε έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από, αυτή την, από αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε πολιτικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις που θα δημιουργήσουν συμμαχίες ε, κατά αυτών των περιορισμών. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι με ενισχύει ιδιαίτερα η κατάσταση των μη κυβερνητικών στην Ρωσία που έχει επιδεινωθεί σημαντικά από το 2012 και έχει άσχημες επιπτώσεις για τα ανεξάρτητα συνδικάτα και τους ακτιβιστές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστικό των θεοκρατικών και πολιταρχικών καθεστώτων στο Καζακστάν. Τα, οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις έχουν συνεχώς ε, μεγαλύτερη πίεση. Οι θρησκευτικές ε, μειονότητες αντιμετωπίζουν συνεχή παρενόχληση και τα δικαιώματά τους καταπατώνται και το Σεπτέμβριο του 2016 είχαμε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα οδηγήσει σε περισσότερη ενίσχυση του κράτους ε, και του έλεγχου του κράτους ε, σε αυτή την περιοχή. Τα πολιτικά κόμματα έχουν περιθωριοποιηθεί. Δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν. Θεωρώ ότι η έκθεση θα μπορούσε να προωθήσει μια αποτελεσματική εφαρμογή της, ε, των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Εκεί όπου η κοινωνία των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινδυνεύουν λόγω της ε, πλήρους χρήσης αυτών των εργαλείων ε, από τους αντιπάλους τους ε, και ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν κενά προστασίας, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών κρατών μελών, των αντιπροσωπιών τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα επιχειρηματικά δικαιώματα επίσης, να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα έναντι αυτών που είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως πάγωμα ξένων λογαριασμών, διεθνές ποινικό δίκαιο και ούτω καθεξής. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά απαραίτητο να θεσπίσουμε μια στρατηγική που θα υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό αποτελεί κομμάτι ενός πολύ σημαντικού συστήματος, του δημοκρατικού συστήματος. Ευχαριστώ. And, uh, two more on the list. Ευχαριστώ. Η Σεσίλ και για να παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ κοίταγα τον τίτλο της παρουσίασης αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της συρρήκνωσης του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες υποανάπτυξη. Βλέπω ότι η μείωση των χώρων αυτών στην ουσία υπάρχει, είναι δεδομένη και στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα της δημοκρατίας η μείωση των χώρων δράσης της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι το θερμόμετρο αυτού το οποίο εμείς ονομάζουμε δημοκρατία. Ας κοιτάξτε τι γίνεται στην Τουρκία και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνω τον κατάλογο. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι πολλαπλοί Υπάρχουν πολιτικά μέσα μείωσης και συρρήκνωσης των χώρων αυτών, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταρρύθμισης νομικών ρυθμίσεων, για τη μείωση του χώρου δράσης. Και δεν επιτρέπει στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν ε, τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ξέρουμε τι γίνεται και στην Ουγγαρία, ξέρουμε τι γίνεται και στον τομέα των πανεπιστημίων στη χώρα αυτή. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσω ακριβώς αυτών των δράσεων των κατασταλτικών δεν μπορούν να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι ε, χρήζουν της βοήθειάς τους. Πολλές φορές οι μηχανισμοί αυτοί είναι έμεση, διακριτικοί και παρόλα αυτά με επιτυχία περιορίζουν την δράση των προσώπων αυτών. Υπάρχουν και νέες μορφές της κοινωνίας των πολιτών, η οποία εκφράζεται όχι μόνο με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως τα λεγόμενα «μουδμόσι του Αγιά, οργανώσεις των νέων, ανεπίσημες, οι οποίες δεν έχουν τα μέσα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούν να δράσουν και να δώσουν τον αγώνα τους. Αυτές οι κινήσεις των πολιτών δεν είναι αναγνωρισμένες νομικά και έχουν δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούν. Είναι νέοι συνήθως, άνεργοι νέοι, οι οποίοι μπορούν να δράσουν για μία εβδομάδα, να διαδηλώνουν, αλλά στο τέλος αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη δράση και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι για λόγους ιδεολογίας βρίσκουν την δύναμη να συνεχίσουν. Συνεπώς λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είναι οι φρουροί της δημοκρατίας. Αυτά είναι τα μέσα λοιπόν και υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι Ξέρουμε ότι στο εσωτερικό, σαν παράδειγμα των χωρών ΑΚΕ, και κλείνω με το θέμα αυτό γιατί μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν, συζητάμε τα θέματα της χρηματοδότησης και μέσα από τις συζητήσεις για τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν χώρες όμως που δεν θέλουν η βοήθεια αυτή να προέλθει από το εξωτερικό, από μια χώρα δηλαδή διαφορετική από τη δική τους. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες οι οποίες δεν το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί χαράζουμε τη τάση που θα ακολουθήσουν οι τρίτες χώρες και με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ε, και θα αντιμετωπίσουν το θέμα της δημόσιας συζήτησης. Όταν υιοθετούμε νομοθεσία ε, για να ε, καταπολεμήσουμε π.χ. την τρομοκρατία. Διάφοροι επιτήτη σε τρίτες χώρες ε, παραποιούν αυτή την νομοθεσία για να ελέγξουν τους όσους διαφωνούν μαζί τους. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν και τελικά δεν επιδιώκουν τους δικούς μας ε, ευαγείς σκοπούς, αλλά αξιοποιούν δική μας νομοθεσία για να επιδιώξουν δικούς τους ε, ε, σκοπούς. Και χαίρομαι που οι ομιλητές στο βήμα και άλλοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το έχουν θίξει το ζήτημα αυτό. Έχουμε νομοθεσία στην Ουγγαρία Έχουμε κοινοβουλευτική έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού από συνάδελφο από το ΕΛΚ, ο οποίος θέλει να ε, ισχύσουν ε, επιπρόσθετα μέτρα ελέγχου για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι η αξιολόγηση των κονδυλίων πολύ συχνά είναι καλύτερη όταν ε, δίδεται η βοήθεια στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όχι σε διμερές επίπεδο τα κονδύλια που δίδουμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις αξιολογούνται επισταμένως, ενώ η διμερής και πολυμερής βοήθεια που δίδεται επισήμως στη χώρα δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και να δούμε ποια συνέχεια δίδεται σε αυτήν μετά και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Αν τελικά δημιουργήσουμε ένα κλίμα που θα μας κάνει να συζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει μια ε, μη κυβερνητική οργάνωση και άπαξ και καταλήξουμε σε αυτό μετά να συζητήσουμε αν θέλουμε να τη χρηματοδοτήσουμε, ε, τότε ουσιαστικά συρρυκνώνουμε εμείς τη δημοκρατία και το ελεύθερο βήμα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Εγώ στο παρελθόν μου έχω εργαστεί ε, σε αναπτυξιακή μη κυβερνητική οργάνωση και νομίζω ότι πολλοί από εσά το ίδιο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει βιώσιμη βιώσιμη δημοκρατία αν δεν υπάρχει βιώσιμη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Γιατί ε, από εκεί προέρχονται όλοι αυτοί οι ηγέτες ε, και επικεφαλής. Και αν το έχετε λησμονήσει, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα παράδειγμα πολύ προφανές, δηλαδή την Νότιο Αφρική. Ε, την Νότιο Αφρική. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ε, είναι μια χώρα η οποία έχει ταλανιστεί ιδιαιτέρως και μετά το Apartheid πέρασε δύσκολα και πριν βεβαίως. Ε, υπάρχει αυτή η κατανόηση του ε, να είμαστε όλοι μαζί ο ένας πλάι στον άλλον, όμως το κόμμα αίσθηση λέει ότι είναι το ίδιο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και δεν υπάρχει λόγος για διαφορετικές φωνές. Εάν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κρίνουμε και θεω ορίσουμε ότι για παράδειγμα η μη κυβερνητική οργάνωση δεν μπορεί να έχει χρηματοδότηση ή μπορεί να έχει χρηματοδότηση επειδή ακριβώς αντίκειται ή συμφωνεί στην TIP-TIP, αυτό συνέβη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ε, τότε ανοίγουμε το κούτι της Πανδώρας, νομίζω ότι θα υπάρξουν διάφοροι κίνδυνοι. Ε, καλωσορίζω τις προτάσεις της εισηγήτριας. Ε, πρέπει να δούμε πώς θα δράσουμε και να έχουμε υπόψη μας ότι για τη χρηστή και καλή διακυβέρνηση σε άλλες περιοχές ε, του κόσμου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια καλά οργανωμένη και κρατεά ε, κοινωνία ε, των πολιτών. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Όλα τα μέλη έχουν εξαντλήσει το χρόνο που ζήτησαν και που τους έχει δοθεί. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να στραφώ στους ομιλητές, στους προσκεκλημένους μας για να υποβάλουν τα σχόλιά τους, να δώσω δύο λεπτά στον κάθε έναν. Ε, κύριε Λάξ, εσείς ε, παρακαλώ είστε πρώτος. Ναι, θα είμαι ε, πολύ σύντομο, ε, συμφωνώ με την κυρία εισηγήτρια. Το οικονομικό βάρος της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα μετατραπεί σε πολιτικό βάρος, σε πολιτικό μοχλό εάν λάβει τις σωστές αποφάσεις. Πολύ συχνά η κρίση μαστίζει τις χώρες αυτές στη Μέση Ανατολή και αλλού και γι' αυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πιο ευέλικτη διπλωματική απάντηση για να αξιοποιήσει ε, τα οικονομικά ωφέλη που με υπομονή αθρίζονται και συσσωρεύονται. Το ζήτημα της αιρεσιμότητας είναι δύσκολο. Ε, δέχομαι στην έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις ενάντια σε όλα τα καθεστώτα που επιβάλλουν περιορισμού στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Μιλούμε για τιμωρητικά μέτρα σε 110-120 χώρε σήμερα. Δεν μπορεί να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Εκεί όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αναπτυξιακά προγράμματα και έργα τα οποία εμποδίζονται από τους περιορισμούς της εκάστοτε κυβέρνησης που στρέφονται προς την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ε, τότε πρέπει να υπάρχει ένας κάποιος συντονισμός ε, ε, και θα πρέπει κάποια δράση να αναλυφθεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση με έμεσο τρόπο θα ήταν μια πολύ διαλλακτική ερεσιμότητα, έμεση ερεσιμότητα έτσι ώστε να προωθήσουμε τα δίκαια μας. Και Βλέπετε ότι οι περιορισμοί, κάποιοι είπαν ότι οι περιορισμοί στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών βαθαίνουν και εντό των κρατών μελών. Στην έκθεση όμω λέω ότι έχουμε πολύ δυναμικά δίκτυα οργανωμένη κοινωνία των πολιτών παντού στον κόσμο που έχουν εμπειρία αντίσταση στην επιβολή αυτών των περιορισμών. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μάθουν από τις οργανώσεις του Μαλή, της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Τινησίας, περιπτώσεις όπου η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ε, με επιτυχία αντιτάχθηκε στους περιορισμούς και τους εξάλληψε. Θα μπορούσαμε και εμείς οι δικοί μας δικαιωτικές χώρες να γίνουν αποδέκτες μάθησης και να αντλήσουν διδάγματα από αυτή την αντίσταση που υπάρχει σε άλλες χώρες του κόσμου. Τώρα, πώς θα έχουμε στήριξη σε μη παραδοσιακές μορφές οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Στην έκθεση μιλώ για την ανάγκη διερεύνησης ε, μορφών στήριξης που δεν θα είναι οικονομικές. Ξέρετε, πολλοί δεν χρειάζονται τις τεράστιες οικονομικές δωρεές που παραδοσιακά ε, συνοδεύουν την, ε, τη βοήθεια. Θέλουν άλλες μορφές στήριξης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διερευνήσει καινοτόμου, τρόπους πολιτικής στήριξης σε τέτοιου είδου κινήματα στο μέλλον και να ξεπεράσει την παραδοσιακή τακτική της παροχής δωρεάς οικονομικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλητρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ναι. Αυτό το ερώτημα της ε, ενίσχυσης της διπλωματικής ε, δράσης είναι ακριβώς ε, αυτό που ήθελα και εγώ να πω και δεν είχα χρόνο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και όχι εύκολο. Αναγνωρίζουμε και αυτό το θέμα της αιρεσιμότητας ως δύσκολο ζήτημα προς εφαρμογή. Νομίζουμε όμως ότι συχνά ακούμε πράγματα σχετικά με το χώρο της κοινωνίας των πολιών και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την σιωπηρή διπλωματία όπως την αποκαλεί, αλλά πάντοτε ανάλογα με τις περιστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλό να γίνει πιο ηχηρή, να μιλά πιο δυνατά και να προστατεύει κάποιες οργανώσεις που κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη διπλωματική της προσέγγιση στον πολιτικό διάλογο να διατηρεί συνεχώς συνάλογο και με την, διάλογο και με την κοινωνία των πολιτών για να γνωρίζει καλά την κατάσταση αυτής της ε, κοινωνίας των πολιτών στις συγκεκριμένες χώρες. Κάποιες φορές ε, γίνονται κάποια επικίνδυνα βήματα για την κοινωνία των πολιτών και είναι πολύ σημαντικό η προσέγγιση αυτή να γίνεται χέρι με χέρι με την κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, αντιπροσωπείες ε, που θα συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών παντού. Και εκεί που υπάρχουν δυσκολίες και εκεί που δεν υπάρχουν, γιατί ο κίνδυνος πάντοτε υφέρπει. Πρέπει να είμαστε προμηθείς, όπως είπατε, λιγότερο επιμηθείς. Αν έχουμε προληπτικά μέτρα, ε, σε χώρες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε προβλήματα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε, κυρία Βέντακ Πλακράις. Ευχαριστώ πολύ. Τρία πολύ σύντομα σχόλια. Το πρώτο έχει να κάνει... Μάλλον και τα τρία έχουν να κάνουν με ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν άμεσα στην Επιτροπή απευθείας σε εμάς ε, για την ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση και τη σχέση της με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κομμάτι των συνθήκων και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο θεματοφύλακα των ε, συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην πραγματικότητα έχει 1,3 δις ε, για την περίοδο 2014-2020, ειδικότερα για να αντιμετωπίσει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όσοι είπατε ως εκπρόσωπος των ειδικών συντεταλμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο που είχα να πω έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Έχουμε φυσικά χρηματοδότηση που δίνεται στην κοινωνία των πολιτών ευρύτερη από το 1,9 2014-2020 που δίνεται για την κοινωνία των πολιτών και, τις, ε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε δύο δις το χρόνο για την κοινωνία των πολιτών και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την ορατότητα και τις βέλτιστες πρακτικές. Συμφωνώ ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που λείπουν και αυτή τη στιγμή πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω σε αυτό το πεδίο. Ε, λίγο πολύ αυτά είναι τα πράγματα που είχα να πω. Το τρίτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην κοινωνία των πολιτών και, της, ε, και την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε αναπτύξει οδικού χάρτες ε, για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους για να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις χώρες. Είναι πέντε χώρες και πάντοτε με χαρά αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα θέματα σε κάθε μία από αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Τερέζα, θέλεις να επανέλθει, να προσθέσεις κάτι? Όχι, απλώς να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω μόνο για την παρουσίαση της κατάστασης, να ευχαριστήσω όσους πήραν μέρος στη συζήτηση. Όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους, και ελπίζω η έκθεση να είναι μια καλή έκθεση η οποία να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα όχι όλες τις πολιτικές θέσεις, αυτό θα είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον τις προτάσεις για την δουλειά την οποία θα πρέπει να κάνουν οι οργανώσεις των πολιτών. Έτσι ώστε να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι σήμερα και να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την δουλειά τους επί τόπου προς την κατεύθυνση τουλάχιστον της δικής μας αντίληψης. Όπως είπε η Τερέσα, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 31η Μαΐου στις 10 το πρωί. Λοιπόν, τελειώσαμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν τώρα δύο προτάσεις εκθέσεις για την Κούβα. Ο Έγγελ είναι ο εισηγητής μας και για τις δύο του δίνω αμέσως το λόγο. Μπορείτε να παρουσιάσετε τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί ο ρόλος μας έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένος εδώ. Είναι μία απλή γνωμοδότηση δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται μόνο της ανάπτυξης, Η πρώτη από τις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνει θέματα αναπτυξιακά σε πολλούς τομείς και αυτό έχει νόημα να εμπλακεί η δική μας επιτροπή. Εμείς δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της αναπτυξιακής δράσης σε τρεις τομείς όπως η Φορεία στη γεωργία, αυτό είναι πολύ σχετικό για μια ανίσο η οποία δεν καλύπτει να καλύψει το σύνολο των αναγκών σε τρόφιμα του πληθυσμού, όπως επίσης και για τις υποδομές του τουρισμού. Ένα άλλο σημαντικό πεδίο είναι η χρήση των φυσικών πόρων για την αηφόρο ανάπτυξη Εδώ χρηματοδοτούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα και κάποια μικρότερα. Και στο τέλος οικονομικές και κοινωνικές οργανώσεις, ένας μεγάλος στόχος, ευρύ στόχος. Ένα από τα θέματα τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, είναι ότι είναι μια χώρα με ε, μέσο εισόδημα άνω του μέσου όρου. Οπότε δεν ε, πρέπει να την χάνει ε, υποστήριξη ε, με τον τρόπο αυτό, αλλά αυτό γίνεται κατ' εξαίρεση μέχρι το 2020. Τώρα αν θα παραταθεί η έκτακτη αυτή ενίσχυση ή θα βρεθούν άλλες λύσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δώσει ο διάλογος στα πλαίσια της νέας συμφωνίας, εφόσον συμφωνήσουμε και εγώ το συστήνω αυτό. Τέλος, για ένα θέμα το οποίο δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη, αλλά έχει σχέση με την Κούβα, κράτος δικαίου, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικές εξελίξεις στην ίσο και το κυβερνητικό σύστημα της χώρας. Ξέρουμε ότι το κυβερνητικό σύστημα δεν αμφισβητείται προς το παρόν, αλλά υπάρχουν εξελίξεις στη χώρα έτσι ώστε να προχωρήσουν ε, σε ελάφρυνση των μορφών διακυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή είναι σε επαφή με την Κούβα, ασχολείται και με τα θέματα του σεβασμού και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο με την Κούβα τα επόμενα χρόνια. και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, από ό,τι γνωρίζω, θα συμφωνήσει με την πρόταση και εγώ συμφωνώ φυσικά και σας συστήνω να την υποστηρίξετε μαζί μου. Ένας έχει ζητήσει το λόγο, ο κύριος Γκουερέρο. Ευχαριστώ. Και εγώ φυσικά είμαι υπέρ του να συμφωνήσουμε με την πρόταση Θα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας σαν κοινοβούλιο στη νέα συμφωνία με την Κούβα και όπως είπε ο κ. Έγγελ, η γνωμοδότηση αυτή είναι μια γνωμοδότηση μικρής εμβέλειας, αλλά συνιστά μια αλλαγή απέναντι στην Κούβα, μια σημαντική αλλαγή, γιατί για πάνω από μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποιες μορφές σχέσεις με την Κούβα, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες και δεν προσανατόλισαν την Κούβα σε κάποιες αλλαγές στον τομέα των ελευθεριών ε, και των κοινωνικών ανοιγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε στην ουσία ε, μια πολυδιάσπαση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κούβα. Και κατά την προεδρία του Μπαρακ Ομπάμα ξέρετε ότι ξεκίνησε το ξεπάγωμα των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κούβα δεν γνωρίζω αν ο πρόεδρος Τραμπ στην παρούσα φάση θα συνεχίσει στην πορεία αυτή. Αλλά τι εξελίξεις επίσης δεν ξέρουμε θα υπάρξουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία συνδέονται με την βοήθεια για την ανάπτυξη που θα πρέπει να βελτιωθούν στην γνωμοδότηση. Εγώ θα παρουσιάσω ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε να δώσουμε σαν παράδειγμα ένα μεγαλύτερο ρόλο στη λογική του φίλου, την λεγόμενη έμφυλη διάσταση, επίσης και ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή τη στιγμή η υπογραφή έτσι και αλλιώς η έκθεση, αυτό προϋποθέτει να ξεκινήσει αμέσως ένας πολιτικός διάλογος για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης ε, σε σχέση με την Ατζέντα 2030. Να κάνω επίσης μια πολύ μικρή διευκρίνηση. Η έκφραση που χρησιμοποιείται ότι η Κούβα θα πρέπει να περάσει σε μια οικονομία της αγοράς. Η έκφραση αυτή δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε το επίθετο κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μια έκθεση, μια έκφραση η οποία συνδυάζει το οικονομικό άνοιγμα αλλά με ισχυρή κοινωνική διάσταση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών καθολικού τύπου προς τον πληθυσμό και ταυτόχρονα κάτι που θα επιτρέψει στη χώρα να πετύχει τους βασικούς οικονομικούς στόχους. Πάντως, το θέμα του Ταμείου, εφόσον συμφωνήσουμε και με το να συνεισφέρουμε εμείς την ενίσχυση τις θέσεις ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έτσι ώστε να αναθεωρηθούν οι σχέσεις με την Κούβα. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, Γκούσμαν. Ευχαριστώ, προ... Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι βεβαίως συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία και στηρίζουμε το διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Κούβας. γιατί έτσι θα σταματήσει αυτό το οποίο ο πρόεδρος Αθνάρ, ο πρωθυπουργός Αθνάρ είχε ξεκινήσει στην εποχή του. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση που βιώνει η Κούβα χωρίς να γίνεται αναφορά στο εμπάργκο των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι στη γνωμοδότηση δεν πρέπει να μιλούμε για τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες στην Κούβα χωρίς να τις εντάσσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με, την ΟΕ, με τον ΟΗΕ είναι στο σημείο 68 ε, η Κούβα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη την ανθρώπινη, δηλαδή υπερτερεί των υπολείπων χωρών της Λατινικής Αμερικής και είναι μέσα από τις πρώτες χώρες της, της Καραϊβικής. Από τις 10 πιο άνισες χώρες ε, στον κόσμο, 6 είναι στη Λατινική Αμερική και η Κούβα δεν είναι μέσα σε αυτές τις 6. Άρα... Άρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε ε, την, ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Κούβα στην ε, συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου, πόσο έχει βοηθήσει περιοχές όπως η Αϊτή, όπως η περιοχή της Σαχάρας, η Ποσαχάρη Αφρική και ούτω καθεξής. Αυτή η γνωμοδότηση ενθαρρύνει τη συμφωνία, ενθαρρύνει το διάλογο και δεν θα πρέπει ε, να λειτουργεί υπονομευτικά και δεν θα πρέπει να είναι μια γνωμοδότηση στην οποία ε, να δίνουμε τάχα μαθήματα στη Κούβα, γιατί ως Ευρώπη πολύ λίγα μαθήματα μπορούμε να διδάξουμε στη Κούβα. Και τι εννοώ, δεν μπορούμε να την παρακινούμε για τη δημιουργία ε, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και περίθελψης όταν έχει το καλύτερο σύστημα υγείας και το καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης σε όλη την Υπηρώτη στη Νότιο Αμερική, τη Λατινική Αμερική. Δεν μπορούμε να τις λέμε να πάει προς μια οικονομία της αγοράς και τον ιδιωτικό τομέα όταν αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που αύξησε τις ανισότητες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην Ισπανία έχουμε 30% παιδική φτώχεια και μαζική ανεργία. Λίγα μαθήματα για οικονομικά μοντέλα θα μπορούμε να δώσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι στην Κούβα. Αυτή η συμφωνία βασίζεται στις συμμετρικές σχέσεις, στο διάλογο μεταξύ των δύο μερών και όχι στην επιβολή του ενός προς τον άλλον και επί του άλλου. Θα πρέπει ο διάλογος να γίνεται με σεβασμό στο κουβανικό λαό και με σεβασμό βεβαίω του κουβανικού λαού προς ε, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ούτε μαθήματα πρέπει να διδάσκουμε, ούτε να επιβάλλουμε τη βούλησή μας. Και η Κούβα θα είχε πολλά να πει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, για τους πρόσφυγες για παράδειγμα και το ποια μεταχείριση επιφυλάσσει η Ευρώπη στους πρόσφυγες ή στους μετανάστες. Άρα ας περιοριστούμε ε, στον σεβασμό και στη συμμετρία μεταξύ των σχέσεών μας. Θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, ε, γραπτά και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Πριν πάμε στο δεύτερο γύρο απαντήσεων με τον Ενρίκε, εκ μέρους της κυρίας Μπετσέρα και συνεισηγήτριας ε, σκιώδους του Άλντε, να πω δύο λόγια. Η κυρία Μπετσέρα προετοιμάζει κάποιες τροπολογίες που θα μας υπεθυμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εργαλείου για τη Δημοκρατία. Είναι ένα εργαλείο για ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ ανάγκη να ενισχυθούν αυτά τα εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε το θεμελιώδη ε, ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Κούβα. Αυτό θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επομένως, αν συμφωνείτε, η κυρία Μπετσέρα θα ετοιμάσει τέτοιου είδους τροπολογίες. Ενρήκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης, αλλά ίσως η Επιτροπή Ανάπτυξης ΔΕΒΕ θα πρέπει να το εξετάσει κάποια στιγμή τη θέση της Κούβας εντός της κοινοβουλευτικής συνέλευσης χωρών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κούβα έχει το καθεστώς του παρατηρητή προς το παρόν και πιστεύω ότι μόλις υπάρξουν και κατοχυρωθούν οι νέες μας σχέσεις με τη χώρα αυτή θα πρέπει να προωθήσουμε έτσι ώστε να προσθεθεί ως μέλος επίσημο ε, τακτικό στην συνέλευση των χωρών ΑΚΕ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Σέφε ε, από τη Ρώμη από την υπηρεσία της Έχετε Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω γιατί έγινε η συζήτηση ήδη στην ΑΦΕΤ και δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα πω είναι ότι θεωρούμε πως αυτή η συμφωνία θα μπορέσει να συνοδεύσει και να επιμηκύνει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη συνεργασία με την Κούβα, γιατί θα αλλάξει τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και θα μας εμπλέξει περισσότερο στην Κούβα. Ε, δεν χρειαζόταν μόνο ο Ομπάμα για να ξεκινήσει αυτό. Η εντολή για τις διαπραγματεύσεις είχε δοθεί δύο χρόνια πριν ξεκινήσει αυτό στη δική του κίνηση προς την Κούβα. Συμφωνούμε όμως ότι αυτή η εμπλοκή είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε και θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα μέλλον που θα βασίζεται σε αυτή την εμπλοκή, την κρίσιμη εμπλοκή. Από αυτή την άποψη λοιπόν καλωσορίζω τις απόψεις που έχουν εκφραστεί σε αυτή την Επιτροπή και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενρία Ταγκέγκα θέλετε να πείτε κάποια λόγια παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ως Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και εμείς καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση και τη δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Άγγελ θεωρούμε ότι πηγαίνει ακριβώς προς τη δική μας κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία που πρέπει να δράξουμε, να την αδράξουμε για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε την Κούβα στην διαδικασία κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης. Όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, δεν πρέπει να κάνουμε κηρύγματα και διαλέξεις, να συνοδεύουμε όλες τις διαδικασίες που ευνοούν την μεταρρύθμιση, να σεβόμαστε τα δικαιώματα και φυσικά τη γνώμη των κουβανών. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε εργαστεί στο επίπεδο της ανάπτυξης με ένα πορτφόλιο 50 εκατομμυρίων το οποίο πηγαίνει προς στρατηγικούς τομείς όπως είπε ο κύριος Έγκελχον. Έχουμε ε, το μηχανισμό ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων μέσω του οποίου έχουμε άμεση επιρροή στις νέες πολιτικές και νόμους στην Κούβα και ενισχύουμε αυτό το στοιχείο του εξυγχρονισμού. Γιατί οι Κουβανοί θέλουν να εξυγχρονιστούν, απλώς δεν θέλουν να τους λένε οι άλλοι τι να κάνουν. Τους αφήνουμε λοιπόν να επιλέξουν οι ίδιοι τι είδους εμπειρογνωμοσύνη θέλουν, σε ποιον τομέα και αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζουμε και με την βιώσιμη ενέργεια, τα προγράμματά μας, βάσει των οποίων επενδύουμε 80 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι αυτή η νέα συμφωνία είναι μια ιδανική πλατφόρμα για περαιτέρω δέσμευση. Για παράδειγμα, μέσα από τα προγράμματα συνεργασίας θα θέλαμε να ξεκινήσουμε και τομεακό διάλογο, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για να μπορέσει κανείς να εμπλακεί και να βρει και νέες ευκαιρίες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μόλις χθε είδα πως η Κουβά έχει το μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή ε, σε όλη την Λατινική Αμερική είναι μεγαλύτερος ε, από το μέσο όρο του ΑΣΑ. Ήθελα απλώς να το τονίσω αυτό. Ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι Κουβανοί είναι έτοιμοι τώρα να παρουσιάσουν ένα νέο ε, νόμο για την αναπτυξιακή συνεργασία και ελπίζουμε ότι με αυτόν θα μπορέσουμε να με τη συνεργασία μας να επιταχύνουμε την έγκριση αυτού του νόμου, ο οποίος εξυγχρονίζει και διευκολύνει τον τρόπο που συνεργαζόμαστε σε επίπεδο ανάπτυξης μαζί τους. Επίσης, όλο και περισσότερο λαμβάνουμε μέρος σε θεματικές γραμμές του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 που τρέχουν σε κοινωνικούς τομείς και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσω είναι ότι οι κουβανοί συμφώνησαν πως Μόλις ε, εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία θα μπορεί προσωρινά να εφαρμοστεί και θα μπορούν και να αποδεχτούν και εθνικά ε, project με θέμα τους ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά μπορεί να φαίνονται μικρά βήματα, αλλά είναι σημαντικά μέσα στα πλαίσια της κατάστασης στην Κούβα. Συνεργαζόμαστε με τους ε, τέρους μας, μεταξύ αυτών και την ΤΕΠ, η οποία προσπαθεί να φτιάξει ένα κονδύλι, έναν τρόπο μεταφοράς των ε, επενδύσεων που χρειάζεται η Κούβα, γιατί τα 50 εκατομμύρια είναι λίγα, δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Έχει εμπλοκή εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα τα σχόλια που ήθελα να κάνω σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Έγγελ. Θέλετε να επανέλθετε, να συνοψίσετε. Ναι, πολύ σύντομα Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για το λόγο κύριο Σολαντιρέρ και Καστιλιάνου. Να πω στους Ισπανούς συναδέλφους ότι το πρόβλημα ενός εισηγητή είναι ότι οι επίσημοι κανόνες είναι τέτοιοι, από τους οποίους εγώ δεν μπορώ να αποστώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μέσω ακριβώς και της διαδικασίας τροπολόγησης, θα μπορέσουμε νομίζω να καλύψουμε ε, την ουσία του θέματος. Εγώ αναγνωρίζω την καλή θέληση όλων και είμαι απόλυτα διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας έτσι ώστε το τελικό έγγραφο να μην είναι μόνο ένα έγγραφο αντιπροσωπευτικό τυπικά, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, κάτι το οποίο θα σας βρίσκει σύμφωνος. Μία μικρή παρατήρηση για τον Ενρίκε. Το τελευταίο θέμα το οποίο έθεσε ο Ενρίκε στα πλαίσια των χωρών ΑΚΕ, της συνεργασίας με τα ΑΚΕ. Αυτό το οποίο προτείνει νομίζω ότι δημιουργεί ένα κίνδυνο να διευρύνουμε δηλαδή ε, τον ρόλο αν θέλετε και τον χώρο εν μιας τέτοιας μικρής περιορισμένης πρότασης. Νομίζω ότι ξεπερνάμε το πλαίσιο της απλής γνωμοδότησης της Επιτροπής μας. Όμως εγώ θα προτιμούσα βέβαια να το κάνουμε και να περάσουμε σε, σε ένα έφετο πλαίσιο ε, στην θέση, στην πρόταση αυτή, είτε εδώ είτε στην Ολομέλεια. Γιατί νομίζω ότι το μέλλον και δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το πώς θα εξελιχθεί το ΑΚΕ σαν οργανισμός αν θέλετε και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει μετά το 2020 στα πλαίσια της λεγόμενης διαφθρωτικής συνεργασίας με τις χώρες ιδιαίτερα της Καραϊβικής. Είναι περιοχές eh, με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα έλεγα, πολύ στενά, όπως ακριβώς και η ΑΦΕΤ. Αν υπάρξει μια συμφωνία συγκεκριμένη με την περιοχή της Καραϊβικής, τότε η Κούβα θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτής της συνολικής συμφωνίας γιατί είναι η πιο μεγάλη χώρα της περιοχής. Αυτό ήθελα να πω. Είμαι στη διάθεσή σας, όπως συνηθίζετε, να εξετάσω τις τροπολογίες σας και να προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη. γιατί το κείμενο το οποίο προτείνω στην παρούσα φάση δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά περιμένω τη συνεισφορά σας μέσω των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η Τετάρτη 26 Απριλίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 30 Μαΐου. Το επόμενο θέμα. Διερευνητική αποστολή στο Τσάδ. Τον Φεβρουάριο μια αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Τσάβ υπό την καθοδήγηση του Ιωακίν Τσέλερ. Νόιζερ, Σαρτζεντίνη και Χέλβανη ήσταν παρόντες. Κύριε Τσέλερ έχετε το λόγο να μας πείτε ακριβώς το τι έγινε στα πλαίσια αυτής της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο τώρα για να δούμε και την γραπτή έκθεση που έχει ετοιμαστεί και να σας τη μοιράσουμε. Εκεί θα δείτε περισσότερα για τις λεπτομέρειες. Ε, ήμουνα επικεφαλής αυτής της αποστολής, τέσσερις ημέρες στο Τσάντ, τρεις μέρες επίσημη αντιπροσωπεία και άλλη μία μέρα ελεύθερη για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τα project της DG ECHO στο Τσάντ, ε, να τα δούμε και να δούμε να τα προσθέσουμε στο πρόγραμμα που είχαμε κατά τα άλλα. Είχαμε πολλούς συνομιλητές από διάφορους τομείς, την κοινωνία των πολιτών. Το Τσάντ απ' έξω δίνει μια εντύπωση μια σταθερής ε, χώρας σε μια σταθή περιοχή. Έχουμε πολλές ε, χώρες εκεί στην περιοχή του Σαχέλ και στην Κεντρική ε, Αφρική που και στην Αραβική Χερσόνησο που είναι σε κρίση, όμως αυτή είναι η εξωτερική εντύπωση. Όταν βλέπει κανείς εσωτερικά πώς λειτουργούν τα πράγματα, εδώ και 25 χρόνια έχουμε τον πρόεδρο Ίντρις Δεμπίτνο, ο οποίος έχει μια μεγάλη οικογένεια, έχει παντρευτεί και έχει κάνει καμιά δεκαριά παιδιά και ασκεί την εξουσία σαν να είναι ο επικεφαλής μιας φυλής ενός κλάν και υπάρχει και μια κλεπτοκρατία, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι φτωχός, όμως η ίδια η οικογένειά του συνεχώς πλουτίζει, γεγονός που οδηγεί σε πολλές εντάσεις ε, στη χώρα. Υπήρξε επίσης ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο τον ε, προσπάθησε να τον ε, ρίξει πριν από 7 χρόνια με τη βοήθεια ε, των γαλλικών ε, στρατευμάτων. Το Τσάντο, όπως λέει και το όνομα, είναι ένα από τα κράτη που γυρνιάζουν με την περιοχή του Τσάντ, η οποία τρομοκρατείται από την Μποκοχαράμ. Έχουμε συζητήσει με τα μέλη της κυβέρνησης. Οι ο Πρωθυπουργός παίζει πολύ σημαντικό ε, ρόλο για την υγεία, για την εκπαίδευση και για την τρομοκρατία που είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες σύμφωνα με τα όσα μας είπε αυτός ασχολείται και με τους ε, φτωχούς ε, και θέλει να το κάνει μέσω της, ε, του, τριπλασιασμού, του τριπλασιασμού του προϋπολογισμού για τη φτώχεια. Μετά όλα αυτά μας κάνανε λίγο να σκεφτούμε. Είχαμε επίσης την ευκαιρία με την υποστήριξη του ΟΗΕ, του, του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, να επισκεφτούμε την περιοχή γύρω από το Τσάντ, να μιλήσουμε εκεί με τον τόπιο πληθυσμό, ο οποίος έχει μια σχετικά καλή ζωή, ασχολείται με τη γεωργία. Τώρα έχουμε πάνω από 100.000 ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να φύγουν από εκείνη την περιοχή λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για περιοχή στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιγόντως ε, ε, το είπαμε σήμερα και για το πρόγραμμα Resilience Αντακτικότητας που είναι πολύ σημαντικό για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε περιοχές σειράξεων γιατί οι πόροι δεν φτάνουν για όλους, ε, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ε, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτές τις περιοχές εξωτερική βοήθεια γιατί δεν υπάρχουν ε, υποδομές μεταφορικές για να έλθουν τα τα αγαθά. Οι οργανώσεις ε, στο πεδίο προσπαθούν να μειώσουν λίγο το πρόβλημα. Ε, έκαναν πολλά πράγματα για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καταστάσεις, όμως όπως είπα αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης είναι ένα κομμάτι που, με το οποίο ασχοληθήκαμε. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχουν περαιτέρω γεωργικές εκτάσεις που θα μπορούν να καλλιεργηθούν ώστε να υπάρχει κόσμος που θα βρει εργασία εκεί και να μπορεί να σταθεί στα πόδια του με τις ίδιες του τις δυνάμεις. Για να... Τώρα βέβαια μένει το θέμα της υγείας και της εκπαίδευσης. Ένα άλλο πρόβλημα του Τσάντ είναι ότι ε, πολλοί από τους πολίτες ήταν πολίτες και της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, έπρεπε να μείνουν εκεί. Ε, πάνω από 25.000 ε, ε, άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να φύγουν από την κεντροαφρικανική δημοκρατία και έχουν πλήρη δικαιώματα ως πολίτες του Τσάντ, μπορούν να δουλέψουν, να έχουν στέγαση και να ασχοληθούν με την επιβίωσή τους, όμως μέχρι τώρα οι διοικητικέ αρχές και κυβερνητικές αρχές δεν τους έχουν δώσει τα απαραίτητα έγγραφα ακόμα. Ζούνε και σε προσωρινούς καταβλισμούς ε, και ε, πολλές φορές εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα πορνείας, ε, διαφθοράς, υπάρχουν τέτοιες διαμαρτυρίες. Εδώ ακριβώς το κράτος αρνείται να παρέμβει και να διοικήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάρα πολλά χρήματα στο Τσάντ για την εξασφάλιση των συνόρων. Βέβαια, επί τόπου ε, φαίνεται ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις, διότι οι συνοριοφύλακες ε, ε, έχουν ε, πρόσβαση στο Καμερούν, στην Ιγυρία ε, και θέλουν να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο μεγάλο σύστημα συναριακής φυλακής. Όμως υπάρχει μια νομαδική μορφή ζωής εκεί στην περιοχή και αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα περιοριστεί πολύ από το πολύ Μαρεγκούρι που είναι μια φυλή στην Νιγηρία θα έχουν πρόβλημα να απολύσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, ε, οι στρατιώτες ε, δεν πληρώνονται καλά. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ε, τα βλέπουν τελείως διαφορετικά οι ντόπιοι για την δημιουργία δυνάμεων ασφαλείας, κυρίως αστυνομίας, Έχουμε δώσει μεγάλη υποστήριξη. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις, ε, όμως ε, παρόλο που είναι έτοιμα τα κτίρια, η εκπαίδευση των αστυνομικών δεν μπόρεσε να ξεκινήσει. Δεν υπάρχει αυτή η βάση εκπαιδευτική και οι αξιώματούχοι μας είπαν ότι δεν έχουν καθόλου χώρους ε, για να κάνουν ασκήσεις σκοποβολής, δεν έχουν χώρους για να κάνουν ε, ασκήσεις ε, παρόλο που έχει δοθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να αντιμετωπιστεί το εμπόριο όμπλων εκεί. Γενικά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διάσπαση και σε επίπεδο υγείας των δυνάμεων. Ε, υπάρχει κάποια νοσοκομεία τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παιδιά. Ε, όμως αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, ε, γιατί δεν αντιμετωπίζονται οι ανάγκες επαρκώς. Πολύ συχνά επίσης το πρόβλημα είναι όχι ο υποσυτισμός των παιδιών αυτών, αλλά οι παραδοσιακοί τρόποι ε, που χρησιμοποιούνται για να γεννηθούν τα παιδιά αυτά, ε, δηλαδή δεν μπορεί να τραφεί μια γυναίκα ε, τρεις μήνες πριν γεννήσει το παιδί και όταν βγαίνει το μωρό είναι πολύ ε, μικρό και είναι και υποσυτισμένο όταν γεννιέται. Άρα εξ αρχής έχει πολύ μικρές πιθανότητες ε, να επιβιώσει. Επίσης, το ίδιο το κράτος έχει φαλυρίσει. παρόλα που έχει πρώτες ύλες, ε, πετρέλαιο και αέριο, είχε κάποια συμβάσεις με την ExxonMobil για πολλά ε, χρόνια. Μετά ε, τον πήρε η Γκλένκο και ζήτησε προκαταβολές ε, από το κράτος. Τώρα έχουν πέσει τιμές πάρα πολύ και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των προκαταβολών και ε, των ε, κερδών αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χρήματα στον κρατικό κορβανά και να έχει φαλυρίσει το κράτος εκ των πραγμάτων, να μην μπορεί να εκπληρώσει τις λειτουργίες του. Η κατάσταση εκεί, ε, στις γύρω χώρες επίσης, έχει δώσει μια θέση κλειδί στο Τσάντ λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Από την άλλη, ε, θα μπορούσε να χάσει την σταθερότητά του και να γίνει ασταθές, ε, όπως βλέπουμε και στις άλλες χώρες που, το, που γυτνιάζουν με αυτό η κατάσταση εκεί επιδεινωθεί, θα μπορούσε και αυτό να αποσταθεροποιηθεί. Άρα είναι σημαντικό από τη μία να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο ίδιο το Τσάντ, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πώς η κυβέρνηση, ο πρόεδρος, το κοινοβούλιο και οι περιφερειακές αρχές ασκούν τα καθήκοντά τους και όταν ε, υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση του ντόπιου πληθυσμού. Επίσης, ένα θέμα που θέλω να, να θέσω είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή ε, Αντιπροσωπεία, η πρέσβυρα Ιονέτα, η οποία από την αρχή είπε, ε, φρόντισε ώστε να έχουμε ένα πυκνό πρόγραμμα θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί μπόρεσε να μας ε, δώσει όλες τις πληροφορίες που θέλαμε και μας ε, συνόδεψε ε, πολύ καλά σε όλη αυτή την αποστολή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πω ότι αυτά που μας είπε ο Γιώχημ ήταν πολύ σημαντικά. Μόνο ένα τεχνικό σχόλιο μείναμε μία μέρα παραπάνω και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για αυτά που κάναμε. Για μένα ε, πάντοτε όταν έχουμε δύο μόνο μέρες για μια τέτοια αποστολή είναι ε, πρόβλημα. Θα πρέπει κανείς λοιπόν να σκεφτεί ε, αν θα ήταν καλό να επιμικρύνουμε αυτές τις αποστολές. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του λοιμού της καταστροφής ε, στα βόρεια της Νιγηρίας ε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ε, μεγάλα κομμάτια στο Τσάντο όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω του Μπόκο και η κατάσταση εκεί να μην έχει γίνει καλύτερη γιατί είναι τώρα σε στρατόπεδα δεν θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους θέλουν να μείνουν εκεί στα στρατόπεδα γιατί στις αρχικές περιοχές από όπου προέρχονται η κατάσταση έχει γίνει πολύ ε, πιο δύσκολη. Έχει ε, η περιοχή αυτή αφαιθεί στη μοίρα της. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την κυβέρνηση για να μπορέσει να φροντίσει για αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό ε, ισχύει και για την πάταξη της τρομοκρατίας, ε, γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να κλείσετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Κάποιοι από αυτούς που συναντήσαμε είναι εκτοπισμένοι, είναι αλληλείς, είναι γεωργοί ε, είναι κτηνοτρόφοι και πρέπει να επιστρέψουν στις περιοχές από όπου έχουν προέλθει γιατί έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και προοπτικές στη ζωή. Ένα μεγάλο τμήμα του Τσάδ θεωρείται όμως ε, δυστυχώς σαν ε, χώρος δράσης πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Μπόκο Χαράμ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας Αλλιώς θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες ζωής και εκεί υπάρχει μια σαφής έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων των τοπικών αρχών. Οπότε επανερχόμεθα στα γνωστά αυτά προγράμματα βελτίωσης της ανθεκτικότητας των τοπικών πληθυσμών έτσι ώστε οι τοπικοί πληθυσμοί και οι νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί να μπορέσουν να βελτιώσουν την τις διαδικασίες επιβίωσής τους. Πάντως μιλάμε για μια τεράστια περιοχή και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πραγματική στρατηγική και μια ισχυρότερη παρέμβαση από αυτήν την οποία μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής που να θέλει το λόγο η κυρία Μπάριος Φερνάντες. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Γεια σας. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτό το μήνυμα. Για την προσέγγιση που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λίμνη του Τσάντα. Θεωρούμε ότι η αποστολή έλαβε χώρα σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται ε, και ε, την αφορούν οι πολλές διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζεται και αυτή η αποστολή εντάσσεται στις λοιπές επισκέψεις και αποστολές του ΟΗΕ και άλλων διεθνών φορέων. Ε, αποκτά μεγαλύτερη ορατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει και οι πολιτικές της για την ανθρωπιστική βοήθεια, για την οικονομική ανάπτυξη, για την ειρήνευση, για όλα αυτά. Η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την επίσκεψη ήταν πολύ σημαντική. Η ευρύτερη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην περιοχή του Τσάτ είναι πολύ σημαντική έγινε μια τοπική δήλωση για την αυθαίρετη κράτηση, κράτηση κάποιων ακτιβιστών φορέων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και έγινε σε συνέχεια της ε, συνεργασίας των ε, μελών του Κοινοβουλίου με τους ακτιβιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα στο Τσάντ και έχει εταιρική σχέση, έχει, δίνει οικονομική στήριξη. Όλα αυτά τα θεωρούμε πολύ σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή, για το, τους κατοίκους στο Τσάντ. Όλα αυτά συνάδουν με το πνεύμα της επίσκεψης. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε. Η Κάρλα Μοντέζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο για να συγχαρεί την ομάδα που οργάνωσε αυτή την κοινοβουλευτική αποστολή, η οποία έλαβε χώρα σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή για ένα θέμα πολύ σημαντικό, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, η περιγραφή της κατάστασης που έγινε για τη χώρα η ανθρωπιστική κατάσταση, η κατάσταση σε σχέση με την ασφάλεια, η ανθρωπιστική καταστροφή ουσιαστικά που μαστίζει τη χώρα λόγω της Μπόκο Χαράμ, όλα αυτά είναι διαπιστώσεις με τις οποίες συμφωνούμε απολύτως και όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε επιτόπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη έχει θεσπίσει ένα σχέδιο οικονομικής στήριξης σημαντικό που ε, θίγει όλους τους τομείς και όλα τα θέματα που ε, τόνισε ο εισηγητής. Έχουμε σημαντικούς εταίρους και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της επισητιστικής επάρκειας, της, ε, του υποσυτισμού, της ανθεκτικότητας του, προ... του πληθυσμού στην ανέχεια στην ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ε, στις χώρες που το χρειάζονται. Και ε, σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την ασφάλεια. Είναι απολύτως προφανές ότι δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι οι αρχές ε, αυτή τη στιγμή δίνουν το βάρος στο θέμα της ασφάλειας και της ανάπτυξης και τις οικονομικές προσπάθειες τις κατευθύνουν προς την ασφάλεια γιατί οι δαπάνες δεσμεύονται εντός του εθνικού προϋπολογισμού για να κατευθυνθούν προς την ασφάλεια και υπάρχει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί η στήριξη του κράτους στο αμυντικό του σκέλος. Άρα ε, μας ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες. Ξέρετε ότι ο αρμόδιος επίτροπος έκανε επίσκεψη μαζί με τον Jean-Marie Leguin, το σχετικό Γάλλο ε, αρμόδιο υπουργό μετά την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό ήταν μια ευκαιρία μεταγενέστερη να τονιστεί για άλλη μια φορά η σημασία που ε, προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών στις εγγυήσεις για την ελεύθερη ύπαρξη διαδηλώσεων, για το δικαίωμα του εκφράζεστε, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις αυθαίρετες συλλήψεις που διενεργούνται αυτή τη στιγμή. δείχνουμε την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας και επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιπρέσθετη οικονομική στήριξη 5 εκατομμυρίων ευρώ έτσι ώστε οι κάτοικοι του Τσάντ να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που απορρέει από την οικονομική και κοινωνική κρίση και που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δράση της Μπόκο Χαράμ και τονίζουμε την ανάγκη για την ύπαρξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεων στον οικονομικό, δημοσιονομικό και φορολογικό τομέα για να κινητοποιηθούν περισσότερο οι ίδιοι οι εγχώροι πόροι που είναι διαθέσιμοι μέσα στη χώρα. Πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η κατάσταση της δικαιοσύνης και η εύρυθμη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας. Η οικονομική στήριξη λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά, ε, η στήριξη αυτή στρέφεται προς όλα τα θέματα, προς όλους τους κλάδους, όλους τους βασικούς τομείς που ε, και η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αναδείξει. Χαίρομαι λοιπόν διότι μαθαίνω ότι πράγματι είχαμε τη στήριξη, είχατε εσείς τη στήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αντιπροσωπεία δούλεψε για να είναι πολύ ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα τους διαβιβάσουμε τα συγχαρητήρια τα δικά σας, των εισηγητών σας και σας ευχαριστούμε εκ μέρου τους για τα συγχαρητήρια που δίνετε στους επικεφαλείς των αποστολών και όλο το προσωπικό που απασχολήθηκε για να ε, λάβει χώρα η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τόσο πετυχημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτά προς το παρόν ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσέλερ, έχετε κάτι να προσθέσετε, όχι. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, όλα έχουν υποθεί σε ό,τι με αφορά. Δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, τα λόγια του Νόρμπερτ. Είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ λίγες οι δύο μέρες για μια διερευνητική αποστολή, εξαιρετικά λίγες και χάρη στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσαμε να μείνουμε άλλη μια μέρα και μπορέσαμε να ε, αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα, να συναντηθούμε με εταίρους ε, με τους οποίους μπορέσαμε να συνομιλήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να είναι και κανόνας εφεξής. Ως προς τα συμπεράσματα που βγήκαν για τις δυσκολίες, πώς μπορεί κανείς να δράσει ενάντια στις δικές του αρχές όταν η κυβέρνηση αφήνει τον κόσμο μόνο του. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, άρα πρέπει εμείς να έρθουμε να καλύψουμε αυτό το κενό και να δώσουμε την εντύπωση ε, στους ανθρώπους ότι τους βοηθούμε και είμαστε παρόντες. Λοιπόν, πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας της συνεδρίασης. Έχετε κάτι υπό τα διάφορα? Όχι, καλώς. Επόμενη συνεδρίαση 3 Μαΐου στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ, κυρίως το πέρας της συνεδρίασης.